Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας αρχίσουμε την ε, ακρόασή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμότατα εξ ονόματος και της κυρίας Βαλεάν, μαζί με την κυρία Βαλεάν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, καθότι πρόκειται για κοινή ακρόαση των δύο επιτροπών μας. Είναι η Επιτροπή Ένβη Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Με θέμα να ε, επαληθεύσουμε κατά πόσο ο προϋπολογισμός συνάδει και είναι συμμορφωμένος με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση της συμβατότητας των ε, σημερινών προϋπολογισμών και σίγουρα και των επομένων. Διότι αυτό τον καιρό προετοιμάζουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020. Συμβατότητα με το κλίμα λοιπόν. Στόχος μας δεν είναι να συζητήσουμε την κλιματική πολιτική, αλλά να εντοπίσουμε τις δαπάνες και τη δέσμευσή τους, δαπάνες για την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμησή της και να αξιολογήσουμε κατά πόσο έχει πληρωθεί ο στόχος του 20%. Αυτά θα συζητήσουμε λοιπόν, καθώς επίσης και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Η παρούσα ακρόαση απαρτίζεται από τρία πάνελ. Το πρώτο θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιση των στόχων ε, της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα. Το δεύτερο πάνελ θα αξιολογήσει το πόσο έχει ενσωματωθεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ε, περίοδου 2014-2020. Και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για τις, οριότητε ε, τις ζώντιες προτεραιότητες. Και το τρίτο πάνελ θα ασχοληθεί με το τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε όλες οι δαπάνες του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, προσφέρουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία σύμφωνη με τις κοινέ μας προτεραιότητες. Και το τρίτο πάνελ λοιπόν θα ασχοληθεί με το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή για το 2030. Κάθε ομιλητή θα έχει περίπου ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσει την άποψή του και τα τρία πάνελ θα έχουν συζήτηση με τους βουλευτές και τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρούσα ακρόαση μεταδίδεται σε web streaming στο διαδίκτυο και θα δώσω μέσα το λόγο στην πρόεδρο κυρία Βαλεάν, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Παρακαλώ. Thank uh, uh, um, Σας ευχαριστώ κυρία Αρτουή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμμετέχοντες, σας καλωσορίζω. Μεγάλη χαρά που σας υποδέχομαι εδώ στην ακρόαση. Όπως υπόθηκε, διοργανώνεται η ακρόαση από κοινού με την Επιτροπή Προπολογισμών. Εγώ, η ίδια, εκπροσωπώ ως Προέδρος την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημοσίας Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας μάλλον και Ασφαλείας Τροφίμων. Θέλαμε πολύ να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή αυτή της ακροάσεως διότι ασχολείται με ένα σημαντικό θέμα που εξετάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η κλιματολογική αλλαγή είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας, η αλλαγή του κλίματος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλο τον κόσμο πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να μειώσουν τα συναφή προβλήματα. Κάναμε μεγάλο βήμα προόδου μέσω της Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι στο ύψο των περιστάσεων. Ξέρουμε ότι στηρίζει ο προπολογισμό του στόχου τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το κλίμα. Έχουμε προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, αλλά αυτό που θα συζητήσουμε εδώ είναι αν αρκούν τα χρήματα για τους φιλόδοξους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος επανειλημμένα προειδοποίησε ότι ελοχεύει ένας σοβαρός κίνδυνος να μην έχουμε πλήρη κάλυψη ε, του στόχου του 20% για δαπάνες ε, ε, για το κλίμα και τονίσαμε ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί για να πετύχουμε το στόχο το 2020. Σε αυτά τα πλαίσια, στην ακρόαση θα εντοπίσουμε την κατανομή των δαπανών για την μείωση των συνεπειών ε, της του κλίματος, αν έχουμε ανταποκριθεί στη δέσμευση του, του 20% και πώς θα ανταποκριθούμε σε μελλοντικά προβλήματα. Ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και εύχομαι μια πολύ καλποφόρα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν αφιβάλλω ότι θα είναι πολύ γόνιμη συζήτηση για το κλίμα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Τάραντ, ο οποίος είναι συγητής ε, της ακράσης εξ ονόματος της Επιτροπής στον Προϋπολογισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και εσάς κυρία Βαλεάν που ήρθατε. Ε, question, Για να συζητήσουμε αυτό το θέμα για να δούμε αν είναι επαρκής οι προσπάθειες που καταβάλουμε. Πολλές φορές στην επί τη σχεδιασμού οικονομία, τι γίνεται. Αυτό το οποίο πάθαμε κι εμείς που κάναμε κάποια σχέδια, αλλά αλλάξαν τα πράγματα πάντως. Η ουσία του θέματος παραμένει. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν είναι θέμα του αν επιτελείται η κλιματική αλλαγή, αλλά το κατά πόσον εμείς επιστρατεύουμε το, το, το οπλοστάσιο που έχουμε. Οπότε μπράβο και σε αυτούς που ήρθαν κατόπιν προσκλήσεως για να τα συζητήσουμε εδώ με τα πάνελ. At a point when uh, the odds for uh, the United States of America to change their position Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες να αλλάξει στάση η Αμερική για τη Συμφωνία των Παρισίων. Α, ούτε είχαμε τίποτα μαντάτα από τον Πρόεδρο ή την κυρία Πρόεδρο, αλλά τίποτα α, από πλευρά των ομολόγων της Αμερικής. Ε, γι' αυτό και χρειάζεται εμεί να είμαστε ένας πιο ισχυρό ε, παίκτη να έχουμε επίσης και ένα προπολογισμό που να ταιριάζει στις δεσμεύσεις των Παρισιών. Και μας καθησύχασε με αυτά που είπε στο Στρασβούργο ο πρόεδρος Μακρόν γιατί είπε ξεκάθαρα ότι η χώρα του θα κάνει και τούτο και εκείνο για να πετύχει τους στόχους. Και θέλω να σας τονίσω τα εξής δύο. Πέρασαν μόλις τρία χρόνια και λιγότερο από την θέσπιση του ισχύοντος πολιτούς πλαισίου και ακόμα δεν πετύχαν τους στόχους για το κλίμα. Να, αυτό είναι το ορεκτικό για να επιληφθούν τα μέλη του πάνελ. Τι πήγε στραβά, γιατί δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει και αυτοί που έχουν την εκτελεστική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πήγαν τόσο καλά. Επίσης, όσον αφορά το επόμενο πολιετές πλαίσιο, εκεί έχουμε προτεραιότητες, έχουμε δει τις επιπτώσεις. Επί τη βάση των όσων συζητώνται εδώ και παντού, για να δούμε πώς θα πετύχουμε όσον αφορά τις δεσμεύσεις των Παρισίων. Οπότε θα πρέπει η αισιοδοξία θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένες πράξεις. Να δούμε τώρα και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Δυστυχώς η χώρα μου βρίσκεται στην απότερη περιφέρεια της Ένωσης και φτάνουν μία μέρα αργότερα οι εφημερίδες. Διάβασαν τους χθεσινούς Financial Times σήμερα και ανακάλυψαν ότι ίσως σύμφωνα με το πολιτές πλαίσιο αλλάξαν τα πράγματα και τα βαλτικά κράτη μπορεί να ρηχτούν υπέρ του Νότου. Να, φουσκώνει το κύμα του πανικού λοιπόν όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για μετανάστευση, για το κλίμα. Θεμητά όλα αυτά, αλλά και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν μένουμε μόνο στα λόγια όσον αφορά τη δέσμευση πόρων για το κλίμα. Θα πρέπει να τα βάζουμε στον πληθωρισμό αυτά και κατόπιν θα πρέπει να ελέγχουμε την εκτελεστική εξουσία. Κύριε Συμπρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ σε τρία σημεία για σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πολύ μια στρατηγική. Θα πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά επίσης. Είχαμε την μελέτη του IPCC για τον 1,5 βαθμό θερμοκρασίας για το ταλανό. Τα νησιά Φίτζ θα σας τα εξηγήσω. Στόχος είναι Οκτώβριος του 18 φέτος και στο ένα και στο άλλο μέρος. Και επίσης είχαμε ε, τη συνάντηση του Κατοβίτζε που θα γίνει το Δεκέμβριο πάλι φέτος και αυτό θα είναι ευκαιρία για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Οπότε, σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό η σημερινή κουβέντα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο προπολογισμό. Μπράβο, μπράβο σε όλους όσοι έχουν χρόνο και ενέργεια για να συμμετάσχουν στην αντίθεση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Αρτουή. Σας ευχαριστούμε έτσι όπως πλαισιώσατε στη σημερινή συνάντηση. με αυτή είναι η δουλειά μας. Να ελέγχουμε το πώς οι φιλοδοξίες και το κλίμα θα είναι μόνο κατάλογος καλών προθέσεων και φραστικά σχήματα. Απ, να το το πρώτο πάνελ. Προεδρεύει η κυρία Βάλεαν. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο πάνελ συζητά προκλήσεις και ευκαιρίες για το προπολογισμό υπό το φως των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα. Έχω την τιμή να καλωσορίσω δύο εμπειρογνώμονες που προσεκλήθησαν για το πάνω. Ο κύριος Φίλιπ Ογουέν από την Γενική Διάθεση Κλίμα και η κυρία Μόνικα Καντάστα, επικεφαλής του Τμήματος για το Περιβάλλον και Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Όουεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και την Γενική Διεύθυνση για την ε, δράση φορά του κλίμα για να εξετάσουμε τις προκλήσεις της ευκαιρίες για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης εν ώψη της Συμφωνίας των Παρισίων Ξυλοποίησεως αυτής. Ήταν πολύ καλό που από πλευρά εισηγητού ετέθη το σκηνικό, διότι ένα από τα δύο σημεία που έθιξε θα τα αναφέρω κι εγώ στη σύντομη, αλλά ελπίζω εστιασμένη παρέμβασή μου. Όπως θα γνωρίζετε, η σημερινή συνεδρίαση είναι άκρο επίκαιρη. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μετά το 2020 στις 2 Μαΐου γίνονται πολύ ζωές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αέναες και δεν σταμάτησαν πρόσφατα ούτε το Σαββατοκυριακό. Είχαμε ηλεκτρονικά μηνύματα που πέταγαν δεξιά και αριστερά. Είναι επίκαιρη συζήτηση, είναι επόμενη Δευτέρα ξεκινά μια συνεδρίαση το ΙΣ οπότε ε, αποκτά η συζήτηση διεθνή διάσταση και ό,τι σχετίζεται για με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη χρηματοδότηση των μέτρων για το κλίμα είναι το θέμα της ε, βιώσιμης χρηματοδοτήσεως. Έχουμε το σχέδιο δράσεως από την αρχή Μαρτίου, Έχουμε, είχαμε την εκδήλωση 22 Μαρτίου των εμπλεκομένων υψηλού επίπεδου ε, και τώρα ε, θεσπίζεται η νομοθεσία. Να επενθυμίσω τρει στόχους, βασικούς στόχους της Συμφωνίας των Παρισιάνων. Καταρχάς, η μέση αύξηση θερμοκρασία να παραμείνει κάτω από 2 βαθμού Κελσίου και να γίνουν μεγάλε προσπάθειε να μειωθεί η αύξηση θερμοκρασία στον 1,5 βαθμό Κελσίου, να αυξηθεί η δυνατότητα να προσαρμοστούμε στι αναπόφευκτε αλλαγέ, συνέπειε αλλαγή του κλίματο, όχι μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαίνει και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι οικονομικέ ροέ θα ταιριάζουν με την ε, αντοχή της τεχνολογίας και να μειωθεί η εκπομπή των αερίων μοκυπίου. Όσον αφορά τη μείωση των συνεπειών, τον Οκτώβριο του 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θέλουμε σε όλη την ε, οικονομία να μειώσουμε 40% τα μοκυπίου μαζί με χρήση ανανεωσίμων πηγών ενεργείας και να έχουμε και 27% ε, βελτίωση της απόδοσης και μείωση των εθνικηπίων. Όσον αφορά τη μείωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα πάει η νομοθεσία που αφορά την ανταλλαγή ρήπων, το ETS που είναι 45% της οικονομίας, υιοθετήθηκε και με τη χρήση υγεών, τα σοκομεία και η λογιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται και ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών, δηλαδή πως τα κάτι μέλη αντιμετωπίζουν το υπόλοιπο 55% της οικονομίας για τη μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αν δούμε τομεακά το θέμα, αυτή την εβδομάδα θα εξεταστεί και το θέμα των βαρέων οχημάτων. Οι αρμόδιοι κάνουν τους σχετικούς ελέγχους. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτά εξετάζονται και προωθούνται τα χαρτοφυλάκια από τον συνομοθέτη. Σε κάτι που είπε ο συγητή, για την αύξηση των φιλοδοξιών μα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πιο πέρα για την ενεργειακή απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε για 27% και πρότεινε 30% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω το Κοινοβούλιο έχει ακόμα μεγαλύτερε φιλοδοξίε σχετικά με αυτό Άρα διατηρούμε αυτέ τι φιλοδοξίε. Τώρα, εκτό των τεκτενωμένων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, έχουμε τι τροπολογίε στο Κιγκάλι του πρωτοκόλου του Μοντρεάλ. Θέλουμε να αυξήσουμε τι φιλοδοξίε των στόχων που πετύχουμε το 2020. Η ΚΑΟ, ένα μηχανισμό βασίζεται στην παγκόσμια αγορά. Και τον Απρίλη, στο Λονδίνο, στο IMO, έχουμε τη μείωση 50% μέχρι το 2050, άλλο στόχο. Πολλά συντρέχουν για τη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Για την προσαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε στατηγική από το 2013. Είναι ένα μέσο που αξιολογείται ούτως ώστε να αναλυθούν περαιτέρω δράσεις στο μέλλον, το βραχυπρόθεσμο. Τέλος, για την βιώσιμη χρηματοδότηση. Έχουμε το σχέδιο δράσης της βιώσιμης χρηματοδοτήσεως που θετήθηκε αρχές Μαρτίου. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Τα χρήματα που θα δοθούν. Αυτό ήταν το υπόβαθρο. Μείωση, ε, βιώσιμη χρηματοδότηση και δημοσίευσαμε 14 Φεβρουαρίου μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μακροπρόθεσμο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και εδώ καθίσατε σαφέστατο ότι ο νέο προπολογισμό έπρεπε να καλύψει θέματα όπω η νέα ζήτηση που, για την ασφάλεια ε, και τη σωστή προσέγγιση και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την μείωση τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην όλη προσπάθεια, όπω λαμβάνεται υπόψη. Και πρέπει να δούμε οικονομίε και την αποδοτική επίτευξη των προτεραιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο και άλλων προβλημάτων θα πρέπει να πολεμήσουμε σκληρά, ώστε η δράση για το κλίμα και συναφεί δαπάνε να έχουν προτεραιότητα στο πολιτικό προσκήνιο, διότι υπάρχουν άλλε στρατηγικέ που ανταγωνίζονται αυτήν. Όμω βλέπω ότι υπάρχουν και ευκαιρίε για τον επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως πάντα ήταν επενδυτικό. και σίγουρα θα υπάρξει συνέχιση τη χρηματοδοτής συνοχή, Διάβασα χθε του Financial Times. Ε, δεν διάβασα αυτό που είπατε να μετακινηθούν χρήματα από το βορρά προ τον νότο αλλά σίγουρα θα υπάρξει ανάγκη επενδύσεων μέσω Ταμείου Συνεχής για τη Γεωργία και μέσω έρευνα και καινοτομία και πρέπει να δούμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως επίσης αναπτυξιακή βοήθεια. Κατά την άποψή μου είναι σαφές ότι η επίτευξη των στόχων του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα θα είναι κάτι δαπανηρό. Στην αξιολόγηση συνεπειών που κάναμε για το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, είδαμε ότι χρειάζονται άλλα 189 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από, από μεταξύ του 2021-2030, τεράστιο ποσό, αλλά πολύ μικρό εν συγκρίση με την αξιολόγηση της διεθνής, του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας για τα 12-13 ε, ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν από τώρα μέχρι το 2030 για να πετύχουμε όλους τους στόχους. Λοιπόν, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μόνο του δεν μπορεί να πετύχει τεράστια ποσά. Τι μπορεί να κάνει όμως να χρηματοδοτήσει πιλωτικά προγράμματα, προγράμματα επιδείξεων να δώσει κίνητρα μειώνοντας τον κίνδυνο για τρίτα μέρη, για τον ιδιωτικό τομέα και τους σχετικούς επενδυτές, ε, να προωθήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι διασυνοριακών δράσεων που δεν μπορεί να πετύχει ένα μεμονωμένο πρόγραμμα ή κάθε κάτω μόνο του αν όλος ο προπολογισμό συμμορφωθεί με τις επιταγές της Συμφωνίας των Παρισίων, τότε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θα μπορούσε να είναι λογικό και σωστό και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Πρέπει να δούμε πιο πέρα στο μέλλον τι γίνεται. Ε, έχουμε, έχουμε λοιπόν, κάνουμε διάλογο γίνεται αποτίμηση, θα γίνει η πρώτη αποτίμηση το 2023 σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τις φιλοδοξίες για το κλίμα, έχουμε τρία ερωτήματα θέσουμε φέτος. Πού είμαστε, αμπρός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχουμε καλή ιστορία να διηγηθούμε, πού είναι τα άλλα μέρη, πού θέλουμε να πάμε. Ήδη είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τους φιλόδοξους στόχους, πού θέλουμε να πάμε μακροπρόθεσμα και πώς θα φτάσουμε εκεί που ειμαστε αν τα ευρωπαικη ενωσεω εχουμε καλη θεωρία να διηγηθουμε που ειναι τα αλλα μερη που θελουμε να παμε ηδη ειπα οτι η ευρωπαικη επιτροπη αυξησε τους φιλοδοξους στοχους που θελουμε να παμε μακροπροθεσμα και πως θα φτασουμε εκει που θελουμε Και η έκθεση του IPCC για τον 1,5 βαθμό είναι πολύ βασικό υπό το φως όλων αυτών. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο εκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια στρατηγική για τα μέσα του αιώνα και καλεί το, επόμενο, το πρώτο τρίμηνο το επόμενου έτου να δώσει αυτή τη στρατηγική για τα μισά του αιώνα. Πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και πριν το Κατοβίτσε να είμαστε έτοιμοι, πριν την κόπ του Κατοβίτσε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στην προετοιμασία θα ξεκινήσουν οι δημόσιες διαβουλεύσεις, έχει δρομολογηθεί η δουλειά και έχει προχωρήσει αρκετά. Δοθέντων όλων αυτών της στατικής για τα μέσα του αιώνα και του διαλόγου και το 2023 θα πρέπει να γίνει αποτίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο, όλα αυτά μπορούν να δώσουν κίνητρα να προχωρήσουμε στην καινοτομία και την έρευνα είναι πολύ σημαντικό, διότι τεχνολογίε που απαιτούνται για τα μέσα του αιώνα ακόμα δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν είναι γνωστέ. Άρα πρέπει να επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτού του τομεί. Και αυτό είναι μια ευκαιρία σίγουρα για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Και αυτό θα επανελειφθεί, διότι το 2023 και το 2028 θα γίνει παγκόσμια αποτίμηση και μπορούμε να το επανεξετάσουμε το θέμα. Και πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά θα δούμε και μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση των τρεχών των προγραμμάτων που θα προταθούν τον επόμενο βήμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη καταλήλως όσο θα προωθεί την νομοθεσία μέσω των θεσμικών οργάνων. Να κλείσω αναφερόμενο σε ευκαιρίες και σε προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τώρα την κατάλληλη νομοθεσία με 12 ορίζοντα. Ξέρουμε που πάμε μέχρι το 2030 και θα θέσουμε και μακροπρόθεσμε στατικές, όχι νομοθεσία, στατηγικέ οράματα για τα μέσα του αιώνα. Δεν είναι μόνο νέο πλαίσιο, για μα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο και θα δημιουργηθεί και ασφάλεια για τι επενδύσει επιχειρήσει και θα προωθηθεί καινοτομιακή έρευνα που απαιτούνται. Σήμερα ε, έχουμε νέε τεχνολογίε και αυξάνεται το τρόπο η ασφάλεια των επενδύσεων. Και είναι επενδυτικό ο του Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μπορεί να δώσει κίνητρο να μειώσει τον κίνδυνο για τα τρίτα μέρη και μπορεί να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία πέραν αυτών. Με βιώσιμο πολιτικό ενδιαφέρον, και είναι τεράστιο αυτό, και βιώσιμη χρηματοδότηση, όλα αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν την όλη εξίσωση. Υπάρχουν κάποιε προκλήσει στον ορίζοντα που διαφαίνονται. Αναφυσβήτητα τα ποσά που εμπλέκονται για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν θα αρκούν για να καλυφθούν όλε οι προκλήσει μα. Και όπω προανέφερα, νομίζω ότι επίση αντιμετωπίζουμε και την αυξανόμενο πολιτικό προβληματισμό για την ανάγκη για κλιματολογική δράση. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει η ασφάλεια, η άμυνα, η μετανάστευση. Υπάρχουν άλλα περιβαλλοντικά θέματα μαζί με άλλα κοινωνικά. Και το κλίμα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα και προτεραιότητα εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω και διεθνώ είναι πολύ σημαντικό διότι έτσι εξασφαλίζουμε τι οικονομικέ ροέ που απαιτούνται από τα διάφορα σχετικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά Μονίκα Σακάστα. Η κυρία από την τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Touch today is ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μια επισκόπηση θα προσπαθήσω να ε, σας δώσω για το τι έχει κάνει η τράπεζά μας αυτό το τομέα ε, και μετά θα μιλήσω για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, γιατί αυτό μου ζητήθηκε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βασικούς στόχους που υποστηρίζουμε και η κλιματική δράση είναι ένας από αυτούς, σαφέστατα και προτεραιότητας. Έχουμε πάρα πολύ σαφή στόχο που συνδέεται με την υποστήριξή μας για τη δράση υπέρ του, τμήματο, του κλίματος. Ε, είναι στο 25% η αύξηση του συνολικού χαρτοφυλακίου για τη δανειοδότηση και την υποστήριξη αναπτυσσομένων ε, χωρών. Και μέχρι το 2020 θα αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση, είπαμε, 25%. Οι στόχοι αυτοί παίζουν ρόλο λοιπόν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ρόλο στην ε, συγκέντρωση της προσοχής ενός ιδρύματος και θεσμικού όργανου όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι αυξημένη η φιλοδοξία λοιπόν για ε, τη χρηματοδότηση από τη θηρίδα ε, χρηματοδότησης καινοτομία ε, των υποδομών. Έχουμε λοιπόν στόχους. Κάθε χρόνο τους καλύπτουμε. Τους καλύπτουμε. Από το 2017 μπορώ να σας πω ότι η χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής ήταν 18,9 και τώρα κλείνει ο τελικός λογιστικός έλεγχος ε, κρεμούν ακόμα, αλλά είναι 19,4 δισεκατομμύρια, άρα 28% ε, του συνόλου της χρηματοδότησης και 2,5 δισεκατομμύρια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι γύρω στο 40% της χρηματοδότησης, της δανειοδότησης μάλλον χωρών αναπτυσσομένων. Φυσικά έχουμε καλύψει τους στόχους. Κάτι άλλο που έχει σημασία και ενδεχομένως να το συζητήσουμε αργότερα είναι το εξή. Πώς κατανέμονται αυτά τα κονδύλια. Έχουμε δυσκολίες στη δανειοδότηση. Ε, μπορούμε να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας σε κάποιες χώρες. Ισχύει αυτό. Πράγματι. Και έχει σημασία εδώ να καταλάβουμε ότι μπορεί να φτάσουμε στους στόχους μας, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και όλοι μαζί να συνεργαστούμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Το κάνουμε και ε, στον τομεακό διάλογο με τους συνομιλητές μας. Δεν αρκούν οι στόχοι από μόνοι Η στρατηγική του κλίματος του 2017 υλοποιείται πλέον πλήρως από την τράπεζα με ε, τα σχέδια δράσης κατά πολέμης κλιματικής αλλαγής. Δεν έχουμε μόνο ποσοτικούς στόχους και μετρήσιμους, αλλά ε, βλέπουμε και μετράμε και τον αντίκτυπο των δράσεών μας και της δανειοδότησής μας επί τόπου και συνεργαζόμαστε ε, με τους ενδιαφερομένους για να δούμε τι σημαίνει η Συμφωνία των Παρισίων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και έργων σε διάφορους τομείς. Όπως μόλις είπε και ο κύριος Όουεν, θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις. για την προσαρμογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε, στην σημερινή πραγματικότητα και είναι μία από τις προκλήσεις αυτές που βλέπουμε δεν αυξάνεται η προσαρμογή και τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία. Και θα έρθω στη συνέχεια σε αυτό τις προκλήσεις και ευκαιρίες. Ε, τρίτος τομέας που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την κλιματική στρατηγική είναι αυτό που κάνουμε και εμείς και είπε και ο κύριος Όουεν ως ανταλλάγματα για κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Πώς θα ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις επενδύσεις αυτό το στοιχείο της κλιματικής αλλαγής διατομεακά. Πώς μπορούμε να βρούμε τις συνέργειες, δεν είναι μόνο κάποια ανταλλάγματα, πώς μπορούν να συνεργάζονται διάφοροι στόχοι πολιτικής και ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις, ποιες επενδύσεις μας βοηθούν να προχωρήσουμε σε διάφορους στόχους. Παράδειγμα, συνέργειες μεταξύ της ατζέντα ε, του θεματολογίου για την κλιματική δράση, για την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν ε, στους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης διάφορες προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των ιδιών πόρων, των υδατίνων πόρων, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με τρόπο συμβατό πάντα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες, συνέργειες και ανταλλάγματα και είναι πολύ σημαντικό αυτό το mainstreaming όπως το ονομάζουμε, η ένταξη ε, αυτής της πολιτικής σε όλες τις πολιτικές. Όχι να υπάρχουν απρός μέσα και εργαλεία ε, όπου να τα εντάσσουμε στην κοστολόγηση των προϊόντων μας όπως είναι η ε, τιμή του διοξιδίου του άνθρακα αλλά να υπάρχει και κανονική εσωτερική δυνατότητα που να, και ικανότητα που να έχουμε αναπτύξει για να καταλάβουμε πώς επηρεάζει κλιματική αλλαγή ε, τους διάφορους κλάδους και πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στην πράξη και να βοηθάμε να ενισχύουμε έργα που έχουν περισσότερο αντίκτυπο στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής ε, διατομέακα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε εστιάσει την τελευταία διετία και πάρα πολύ σημαντικό είναι από τις σημαντικές προκλήσεις προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ε, δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτικές. Θα πρέπει τα επενδυτικά κονδύλια να πηγαίνουν στα σωστά προγράμματα. Και εκεί είναι θέμα ικανοτήτων, ε, περιορισμών αλλά και ευκαιριών. Αυτό είναι ας πούμε κάτι που βλέπουμε ε, με την υποστήριξη από το Συμβουλευτικό Κόμβο και τις ειδικέ ε, πρωτοβουλίες που στοχεύουν προς τα εκεί. Και έχουν ακριβώς ως ομάδα στόχο κάποιες μονάδες ε, που έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση της συμφωνίας. Βλέπε δήμους, κοινότητες, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει το πρόγραμμα Urbis και παγκόσμιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συντονισμό και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς. Θα έχουμε λοιπόν εκεί να διαδραματίσουμε ρόλο υποστηρικτικό ε, στο σχεδιασμό, στην υποστήριξη για καλύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων και τελικά για αύξηση της ε, επένδυσης, της για την κλιματική αλλαγή. Θέλω να επιστρέψω λίγο και να αναφέρω ένα άλλο στοιχείο που χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη ε, για τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν επενδυτικά προγράμματα είναι ε, η εκτίμηση και η διαχείριση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης ε, κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα επεκταθεί σε όλα τα προγράμματα, η διαχείριση. Μέχρι τέλη του 2020 θα υπάρχει παντού αυτό το σύστημα διαχείριση του κλιματικού ελέγχου δεν έχει να κάνει μόνο με το screening και την τακτοποίηση του κινδύνου, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τις λύσεις που χρειάζονται και τους απαραίτητους πόρους. Αυτό εμεί μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε την ε, πραγματογνωμοσύνη και την ε, εμπειρογνωμοσύνη στο συμβουλευτικό κόμβο προ οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αποτανθεί σε εμά. Αυτό τον καιρό συνομιλούμε με ένα κράτος μέλος, αλλά στόχος μας είναι ε, να προχωρήσουμε και με τα άλλα κράτη. Ένα τελευταίο που θέλω να σας αναφέρω είναι το εξής. Ανέκαθεν λέμε ότι ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν πρόκειται να φτάσει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ενδιαφερθούν και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα για μια αηφόρο και βιώσιμη χρηματοδότηση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παίζουν ένα διπλό ρόλο. Έχουμε πραγματογνωμοσύνη για την κινητοποίηση ιδιωτικών κονδυλίων στο κλίμα και μόνο. Αν κοιτάξουμε τους πόρους θα διαπιστώσουμε ότι κινητοποίησαμε επιπλέον κεφάλαιο της τάξεως ε, με μόχλευση τριπλάσια με τετραπλάσια από ε, την αρχική ε, δική μας χρηματοδότηση και σε μικρά προγράμματα επιτόπου αυτό μπορεί να φτάνει και πολλαπλασιασμό επί 23. Είναι τεράστια λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα της μόχλευσης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεκτικό Συνέδριο ε, τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και λογοδοσία δεν πρόκειται ε, να αλλάξουμε τον τρόπο χρηματοδότησης ή κυκλοφορίας των κεφαλαίων ε, μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων αν δεν υπάρχει σαφήνεια και στους ορισμούς και ας πούμε στην έκδοση ομολόγων που εμείς ήμασταν πρωτοπόροι πριν από 11 χρόνια και στην Ουάσιγκτον έχουμε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε λοιπόν ένα ρόλο πρωταγωνιστικό, πρωτοπόρο που δείχνουμε ότι όλα αυτά είναι δυνατά και είναι και αξιόπιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της αγοράς και δημιουργία μιας αγοράς για να ακολουθήσει και η ιδιωτική χρηματοδότηση ε, στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Και γενικότερα στους στόχους της αηφορίας. Θα σταματήσω εδώ και με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας για τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Συνάδελφοι, θέλει κάποιος να διατυπώσει μια ερώτηση προς τους ειδικού μας. Όχι, παρόλα αυτά οι παρατηρήσεις που κάνατε και οι δύο είναι πολύ σημαντικές για μας. Και ισχύει αυτό. Έχουμε θεσπίσει νομοθετήματα. Όμως είδαμε ότι έγινε μια μεγάλη στροφή στα οικονομικά και στο επιχειρήν συγκεκριμένα. Είδαμε πώς ελκύσαμε οι δυτικές επενδύσεις. Και τα προγράμματα για το κλίμα πρόκειται να ανταγωνιστούν τις άλλες μας προτεραιότητες. Βέβαια και τελικά θα πρέπει όλα αυτά να είναι αποδοτικά για να υποστηριχτούν. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για το τι χρειάζεται, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, περισσότερη μόχλευση. Να, μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Α, ο κύριος Τάραντα έχει μια ερώτηση. Όχι, όχι. Πρώτα, κύριο Σόλα. Uh, Τελικά ο κύριο Στάρνα παίρνει το λόγο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. έχω εγώ μια ερώτηση προς την ε, ΕΤΕ, διότι διάβασα, όχι, όχι, όχι στο Financial Times, ότι έχετε διαθέσει σημαντικούς πόρους σε μια εταιρεία που ονομάζεται Volkswagen. Αυτό. Στον ισολογισμό σας. Πώς θα καταχωρηθεί ως δράση για το κλίμα ή αλλιώς. Σόλε. Ο Ευχαριστώ για όλα όσα μας παρουσιάσατε. Είναι σαφές ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας για κλίμα και ενέργεια. Επομένως, τελικά θα πρέπει να μπλέκουμε όλοι οι σχετικοί. Και η διοίκηση, η διακυβέρνηση σε κάθε επίπεδο, για τον άνθρακα, για όλα που έχουν σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη. Συνήθως οι περιφέρειες, οι δήμοι έχουν σημαντικό ρόλο. Και σε εκείνο το επίπεδο τα πράγματα διακρίνουν περισσότερη φιλοδοξία. Άρα, ρωτώ, εσείς πώς θεωρείτε ότι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούμε να έχουμε περισσότερη εμπλοκή με τον προϋπολογισμό κίνητρα, περισσότερο να ασχοληθούν τέλο πάντων οι τοπικέ αρχέ. Πώς θα πρέπει να γίνει η δαπάνη, η διάθεση των πόρων. Thank you very much. Now, Mr. Horvath. Ο κύριο Χόρβατ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγιος Χάουαρτ. Mm. Μα είπε για την ευσημότητα στα έργα και προγράμματα και θέλω να το πάω παραπέρα. Με ποιο τρόπο θα είμαστε πιο αποτελεσματική για τις προτάσεις της ΕΤΕΟΥ ώστε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβουμε στο Παρίσι. Και τι γίνεται με άλλους τομείς, τους άλλους τομείς του προπολογισμού πρακτικά. Ευχαριστώ κύριε Ντάλη. Ε, εγώ ευχαριστώ πρόεδρε. Και αλλά και τους ε, εισηγητές μας. Να δούμε από πλευράς περιβάλλοντος. Μια που στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εργάζομαι. Πρόσφατα είχαμε διάφορες προτάσεις, νομοθεσίες, νομοθετήματα για το περιβάλλον και το βασικό πρόβλημα ήταν πώ θα εξασφαλιστεί ότι αυτά τα νομοθετήματα που θεσπίζονται είναι στο ίδιο μήκο κύματο με τι δεσμεύσει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Και τα τρία θεσμικά όργανα, το θέμα είναι αν έχουν αρκετή φιλοδοξία, ούτως ώστε να τα καταφέρουμε. Και να κάνουμε κάτι για την αλλαγή του κλίματος. Νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, και υστερούν οι προσπάθειές μας. Δεν λαμβάνονται τα πιο δόκιμα μέτρα και πρωτοβουλίες. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι για το κλίμα, να είναι πρωτοπόρα, θα πρέπει να αφιερώσουμε πόρους, μια καθαρή οικονομία κλπ και για την περίπτωση το 2020 και αυτά ανεβούν τώρα υπόψη στις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω δύο ερωτήματα, εάν μπορείτε να με διαφωτίσετε. Πρώτα-πρώτα, πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα πρόοδου με την χρηματοδότηση, να πάμε σε βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες, πώς όλα αυτά θα γίνουν πράξη, τι πρωτοβουλίες γίνονται. Άλλη ερώτηση για τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά κυρίω την πράσινη χρηματοδότηση. Και έτσι να γίνει μετάβαση σε μια οικονομία, σε έναν κόσμο με λίγη χρήση άνθρακα και ανθρωπικές οικονομίες. Πάμε τώρα πίσω στους ειδικού μας. Ποιος θέλει να πάει το λόγο πρώτος? Maybe Mr. Owen first, yeah. Ο καθένας έχει το μερτικό του της ερωτήσεως για να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συμπρόεδρε. Και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Εν γέννη απευθύνονται στη συνάδελφό μου τη Μόνικα και στις γνώσεις που έχει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να αναφερθώ σε άλλες στοιχές. Κάποια ερώτηση αφορούσε τα κίνητρα που χορηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Ευρύ το φάσμα της ερώτησης. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια ρυθμιστική, ασφάλεια δικαίων. Υπάρχει νομοθεσία μακροπρόθεσμη μέχρι το 2030, με ένα όραμα και πέρα από αυτή την προθεσμία. Αυτό δίνει κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με αυτό έχουμε διάφορα επενδυτικά ταμεία και πόρους υπάρχουν και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν εγγυήσει ή όχι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουμε ιδιωτική χρηματοδότηση, ενεργειακή απόδοση την χειρίζεται η οχι που μπορουν χρησιμοποιηθουν εχουμε Τράπεζα Επενδύσεων Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό για τιμή των κινδύνων. Ασφάλεια δικαίου, ρυθμιστική ασφάλεια και χορήγηση κινήτρων. Είναι δύο εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε. Άλλη ερώτηση. Πώς μπορεί να συμμετάσχει η τοπική αυτοδίκηση και διάφοροι ντόπιοι φορεί. Ένα πρόγραμμα εμπίπτει στην... είναι το πρόγραμμα Life που εμπίπτει στην αρμοδιότητά μα και εφαρμόζεται σε τόπιο επίπεδο. Συμμετέχουν οι ΜΚΟ και ωφελούνται οι ΜΚΟ και για την προστασία της φύσης και για τα διάφορα προγράμματα για το κλίμα και περιφερειακές αρχές, πόλεις, δήμοι ωφελούνται από το πρόγραμμα και συμμετέχουν. Πρέπει να έχουμε γενικούς στόχους σε ψηλότερο επίπεδο. Βέβαια. Μπορούν όμως και οι ντόπιες αρχές και φορείς να συμμετάσχουν. Έχουμε και το σύμφωνο των δημάρχων, που είναι ένας φορέας που μπορεί να κινηθεί για την μείωση των συνεπειών του κλίματος και την προσαρμογή σε αστικό επίπεδο στις αλλαγές του κλίματος. Η ερώτηση της κυρίας Ντάλη πώς μπορούμε να προσανατολίσουμε τον προπολογισμό προς βιώσιμε πρακτικέ και, προϋπολογι... Ε, τεχνικές. Έχουμε ε, το πρόγραμμα 9 που κινείται προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, κάνουμε πρόταση εμείς. Οι συνομοθέτες μπορούν να επηρεάσουν προς αυτή την κατεύθυνση της προτάσει μας. Κατά την άποψή μας πρέπει να πω ότι υπήρξε για την έρευνα και την οτομία και το παρελθόν προσπάθεια να, συμμε... να λαμβάνονται υπόψη πτυχές του κλίματος, οπότε όταν δίνονται χρήματα για έρευνα λαμβάνεται υπόψη και το κλίμα και όλος ο προπολογισμό του Πρακής Ενώσεως υπόκειται σε αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Έτσι θα ξέρουμε κατά πόσο πετυχαίνουμε τους διάφορους στόχους μας με τα χρήματα που διαθέτουμε. Επίσης μιλάμε και για την εφαρμογή των στόχων για το κλίμα και του στόχου ηγετία, όσον αφορά την πράσινη χρηματοδότηση πλευρά κρατών μελών. Είναι πρώιμο το στάδιο. Έχουμε σχέδιο δράση για βιώσιμη χρηματοδότηση. Υιοθετήθηκε αρχέ Μαρτίου. Μου λένε συνάδελφοι ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει την προσέγγιση. Πρέπει να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε. με την πάροδο του χρόνου η προσέγγιση γίνει νομοθεσία, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις ιδέες μας και την νομοθεσία μας στο σχετικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κατάστα. Ευχαριστώ. Για να δω αν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αρχίζω από το τελευταίο το οποίο ανέφερα. Ας σταθούμε μια στιγμή. Συγκεκριμένα πώς συνεργαζόμαστε με τα διάφορα στοιχεία από τις χρηματαγορές και πώς συνεισφέρουν, με ποιο τρόπο. Ας αρχίσουμε από ένα απλό, ας πούμε, παράδειγμα συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας που είναι ε, χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεση. Αυτό είναι το πρώτο ε, σημείο αφετηρίας για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ε, ποιες είναι οι δραστηριότητές μας, ιδιαίτερα στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά και για τη βιομηχανία. Ε, συνεργαζόμαστε με τους χρηματοοικονομικούς ενδιαμέσους για να καταλάβουν ποιες είναι οι διάφορες δραστηριότητε και τι εκθέσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε φορά ε, για να ε, μπορέσουν οι τράπεζες να εξετάσουν το χαρτοφυλάκιό τους ως σχετικό με την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Επίσης έχουμε και ένα εργαλείο για την ηλεκτρονική εκμάθηση, για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά πρότυπα και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και νομίζω ότι θα το ε, επεκτείνουμε και θα το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο άμεσος σύνδεσμος με τους ενδιαμέσους. Μετά, Υπάρχει ειδικό σχεδιασμό συγκεκριμένων εργαλείων ε, για να ε, προσελκύσουμε επιπλέον ιδιωτικά κονδύλια. Και πάλι αρχίζοντας από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο ε, μπορούμε ας πούμε να αναφέρουμε επένδυση σε κάποια project που έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή με την ενεργειακή απόδοση. Και τι έχουμε διαπιστώσει ότι οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κλάδο ή σε αυτά τα ταμεία, μάλλον η ίδια η παρουσία μας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, δρά ως ε, κίνητρο για να συμμετέχουν και άλλοι. Δίνει κάποια αξιοπιστία και κάποια στιβαρότητα ε, στο όλο υπάρχουν ας πούμε ε, διάφορα ταμεία που είναι σε, σε στρώσεις. Ένα ταμείο ταμείων, άλλα επιμέρους ταμείο που έχουν ε, συγκεντρωθεί ε, οι πιστώσεις των δωρητών, οι υποσχέσεις, η προστασία από απώλειες του πρώτου καιρού λειτουργίας, το first loss κτλ. Όλα αυτά έχουν γίνει και με το Ταμείο για ε, την ενεργειακή απόδοση και κάποια άλλα ταμεία που έχουμε για εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ταμείο ταμείων για τις ανανεώσιμες και τα λοιπά, που έχει έρθει τώρα στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο στάδιο της λειτουργίας και κατάφερε στην πρώτη φάση να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις. 20 πλάσεις ή 30 από την αρχική μας. Αυτά είναι για τα διάφορα μέσα. Ωστόσο, για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος επανέρχομαι σε αυτό που υπόθηκε για ε, το πρόγραμμα δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ε, ορίσει σαφώς την ε, ταξονομία, να ξέρουμε ε, ποια κονδύλια πηγαίνουν πού. Είναι σημαντικό αυτό για να μετριαστούν οι ζημίες. Ε, συνεργαζόμαστε ε, με τις μονάδες ε, στις οποίες ε, έχουμε τη, τη δράση μας για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε. Έγινε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη Volkswagen. Εντάξει, εκεί πρόκειται για απάτη, για εξαπάτηση. Και ε, πραγματικά ε, αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εργαστεί και έχει διαθετήσει όλα τα μέτρα ε, για ε, την καταπολέμηση της απάτης. Έχουν αποπληρωθεί τα δάνεια προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει σταματήσει η χορήγηση δανειών προς τη Volkswagen και έχει πάρει το δρόμο της η υπόθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρόκειται γενικά για θέματα κλιματικής αλλαγής. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρόλο των τοπικών ε, κοινωνιών και γενικότερα των διαφόρων ενδιαφερομένων, έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο πραγματικά θεμελιώδη. Οι πολίτε, οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι κοινότητες, γενή, η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό γίνεται διεθνώς και γίνεται και αισθητό διεθνώ. Στην COP23 κάποιο είπε ότι απουσίαζαν οι πολιτείες. ήταν παρούσες όμως πόλεις, πολιτείες. Ε, represent... ε, ο ιδιωτικό τομέα κλπ. Ήταν παρούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, ίσως όχι σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά οι τοπικές κοινωνίες βεβαίως και συμμετέχουν. Και σε αυτό το επίπεδο επίσης πρέπει να είναι ε, παρούσα η χρηματοδότηση ή δανειοδότηση. Ε, το τονίζω πάντα αυτό. Και πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Σύμφωνο των Δημάρχων και με τις διάφορες εταιρικέ σχέσεις και σχήματα που έχουν και με εμά, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, με την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα ιδρύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συνεργασία λοιπόν για να δούμε και ποιοι είναι οι διακριτή ρόλοι του καθενός και η συνεργασία. Γιατί δεν είναι όλες οι τράπεζες ίδιες ή όλοι οι οργανισμοί Άλλοι είναι για το διάλογο πολιτικής, άλλοι είναι για τη χρηματοδότηση, για τη δανειοδότηση, όπως είμαστε εμείς, αναπτύσσουμε προγράμματα επενδυτικά, τα προωθούμε και τα εκτελούμε στη συνέχεια. Μαζί, πάντα και κινητοποιώντας ε, τον ιδιωτικό τομέα. Έγινε κάποιους λόγους για όρους και προϋποθέσεις, λεγόμενη αιρεσιμότητα. Για να πετύχουμε ε, στην ανάπτυξη αυτών των χαρτοφυλακίων μας για την κλιματική αλλαγή, αυτό δεν έγινε με όρους και προϋποθέσεις, αλλά με διάλογο και με κάποιες ε, δρομολογήσεις κάποιων έργων ε, στοχευμένων, ε, με κοινούς κανονισμούς, μάλλον με κοινούς ορισμούς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εκεί παίζουν ρόλο οι στόχοι, δεν αρκεί να, να θέτεις στόχους για να δραστηριοποιούνται εκείνοι που χαράσουν τα επενδυτικά προγράμματα ε, officers τους ε, λέμε εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι στελέχη που καταρτίζουν διάφορα προγράμματα ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζεται μόνο γενικό στόχο, αλλά συγκεκριμένο πρόγραμμα με πολύ αξιόπιστο τρόπο. Και όλα στα στοιχεία για το κλίμα ε, λογιστικό έλεγχο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Είμαστε ο μόνος οργανισμός που υφίσταται λογιστικό έλεγχο σε όλα αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά. Για το μέλλον τώρα αναλύουμε όλα τα χαρτοφυλάκια για να δούμε και ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες παντού σε όλα τα μέρη της γης και σε όλους τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας. Και ένα σημείο που θα πρέπει να εντοπίσουμε είναι ακριβώς ποιες αδυναμίες έχουμε, πού δεν προσαρμοζόμαστε, ε, έχουμε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο χρηματοδοτικό μέσο, κάποια συμβουλευτική δραστηριότητα που μας έχει διαφύγει. Εκεί είναι λοιπόν τα σημαντικά στοιχεία. υποστήριξη ακριβώς νέων τρόπων ε, λειτουργίας. Χρειάζεται νέα τακτική, νέα συμπεριφορά, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και πάλι εκεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντική. Στην αρχή είναι μικρά τα έργα, δύσκολα στην εκκίνησή τους, αλλά σιγά σιγά ε, μπαίνουμε σε μια νέα λογική και τώρα χρειαζόμαστε κονδύλια σε ένα τομέα που, που μέχρι σήμερα ε, χρηματοδοτείται από επιδοτήσεις και μόνο και όχι από δάνεια. Και όταν βλέπει και η αγορά ότι πιάνουν τόπο, έχουν νόημα αυτά που κάνουμε, κινητοποιούνται και τα ιδιωτικά κεφάλαια και έρχονται και ιδιωτικέ επενδύσει. Αυτό είναι το μοντέλο μας και ελπίζω να επεκταθεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις. Uh, Όχι ακόμα. Ο πρόεδρος Αρτουή θέλει να θέσει ερώτηση. Απευθυνόμαστε στο πάνελ. Ο κ. Αχτουή. Μάλιστα. Εκφράζω την έκπληξή μου. Διότι δεν αναφερθήκατε σε νέους ιδίους πόρους ενδεχομένους. Όταν αναφερόμαστε στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναφερόμαστε και σε νέους ιδίους πόρους. Και κυρία μου, αναφερθήκατε στο μοχλό που μπορεί να πείσει τους διάφορους φορείς. Η φορολόγηση δεν θα μπορούσε να είναι κάτι που μπορεί να προσανατολίσει, προσανατολίσει συγγνώμη, τη συμπεριφορά. Ένας φόρος άνθρακα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας για μια αγορά άνθρακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με που θα καλύπτει το μειόμορφα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα μπορούσε να είναι μοχλός που χρειαζόμαστε. Εξάλλου, ποια είναι η άποψή σα, όσον αφορά την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ φορολόγησης επί των καυσίμων σε εθνική κλίμακα με τη φορολόγηση στις διεθνείς μεταφορές. Θεωρείτε ότι θα μπορούμε να παράσουμε από φορολόγηση τα καύσιμα των αεροσκαφών και των πλοίων στο διεθνές εμπόριο, ΕΣΑΗ, e, ενώ στις μεταφορές τις εγκύτερες υπάρχει φορολόγηση που βαρύνει τα καύσιμα. Κάναμε άμεσο συσχετισμό μεταξύ του επομένου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και της δημιουργίας των νέων ιδίων πόρων δημιουργήσαμε πολύ στενή σχέση μεταξύ των δύο. Δεν θεωρείτε ότι όσον αφορά την σωστή συμπεριφορά που επιθυμείτε η φορολόγηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοχλό, μια κινητήρια δύναμη, ένα κίνητρο για να αλλάξουν οι συμπεριφορές. Απάντηση. Σε όλα τα μέλη του πάνελ πρέπει να απευθύνουμε τις ερωτήσεις. Ο κύριος Όουεν μπορεί να απαντήσει. Σύντομα να σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Είναι θεμητό να πούμε ότι στις δεκα... στην ανακοίνωση της 14ης Φεβρουαρίου είχαμε συζητήσει διάφορες, διάφορους ίδιους πόρους που αφορούσε και το σύστημα ανταλλαγής ε, ε, ρήπων, ΦΠΑ, ε, μία βάση για φορολόγηση επιχειρήσεων και τον φόρο επί των κεντρικών τραπεζών που μπορεί να εκδίδουν χρήμα. Όλα αυτά συζητήθηκαν εκτενώς. Πράγματι, με την απόσυση του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους νέους τομείς άμυνα, ασφάλεια, μετανάστευση που καλύπτονται, υποτίθεται και φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση αν θέλουμε να κατήσουμε τα επίπεδα δαπανών που απαιτούνται. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις των λεπτομεριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ιδίους πόρους. Σε καμία εβδομάδα ξέρουμε όλοι που βρισκόμαστε. Τα δύο θέματα που αναφέρατε, τον φόρο του άνθρακα, το εξετάσαμε επιμακρών στις υπηρεσίες. Υπάρχουν προβλήματα όμως όσον αφορά τη μεθοδολογία, πώς μπορεί να εφαρμοστεί σωστά. Πώς μπορείς να καθορίσεις το περιεχόμενο άνθρακα που εισέρχεται χάλιβα από μια χώρα, χάλιβα από άλλη χώρα, κράματα από χάλιβα, δύσκολο. Ποτέ δεν είμαστε υπέρ της φορολόγησης με βάση τον άνθρακα ε, στα σύνορα, κυρίως όταν έχουμε σύστημα ανταλλαγή ε, εκπομπών εντός της α, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορολόγηση επί καυσίμων έχει συζητηθεί όπως και γενικότερα φορολογικά θέματα. Δεν έτυχε υποστήριξη σε αυτή η φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο σχετισμό με τις διεθνεί μεταφορές κάπου προχώρησε, αλλά χρειάζεται η αλλαγή διεθνών συμβάσεων. Η αεροπορία διέπεται, οι αερομεταφορές από τη σύμβαση του Σικάγου, από ό,τι θυμάμαι. Άρα, χρειάζονται διεθνείς συμφωνίες για να γίνουν αλλαγέ. και χρειάζεται και συζήτηση με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία. Λοιπόν, επίσης πρέπει να ληφθεί απόφαση ομόφωνα στο Συμβούλιο για τη φορολόγηση και αυτό είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Σίγουρα, σίγουρα λέει και ο Σαχτουή. Αλλά αν ξεκινήσετε από εκεί, από αυτή την άποψη, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει κάποτε η συζήτηση να ξεκινήσει ενώπιον της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης. Δεν μιλάω για τη φορολόγηση των εταιριών, για φορολόγηση που δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρακα. Στοχεύω τον άνθρακα διότι αυτός βοηθά να σεβαστούμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Και όχι διότι υπάρχουν συμβάσεις ε, απερχιωμένες που κάποια στιγμή λαμβάνοντας υπόψη το ότι αλλάζει ο κόσμος ε, δεν θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τα πάντα από την αρχή. Αν δεν κάνουμε, αν δεν κινηθούμε θα συνεχίσουμε έτσι. Μπορούμε να διακηρύσουμε φιλόδοξους στόχους επί τη ευκαιρία τη συμφωνία των Παρισίων, αλλά δεν θα εφαρμόσουμε τίποτα. Θα διονύζεται εικόνα μιας πολιτικής δύναμης ε, που ε, δείχνει πόσο αδύναμη είναι. Εκτίθεται από την αδυναμία της να δράσει. Κυρία Σκατάστα, όχι, πρόεδρος μάλλον, ο πρόεδρος Μακρόν θα πείσει το Συμβούλιο να προχωρήσει. Το Συμβούλιο μακάρι να εισεκουστείτε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ζητούσαμε τα έσοδα από το ETS να χρησιμοποιηθούν για το περιβάλλον και σχετικά προγράμματα. Το Συμβούλιο όμως ε, είναι δύσκολο με τα θέματα του προπολογισμού είναι πολύ κτητικό. Ελπίζουμε κάτι να αλλάξει. Θέλετε κι εσείς να λάβετε τον λόγο. Κυρία Σκατάστα, θέλετε να μιλήσετε. Θα απαντήσω γαλλιστή. Ετέθη γαλλικά το ερώτημα. Διαπιστώ ότι μπορώ να σας απαντήσω ως ηθικός. Αλλά ξέρω αν θα είναι η θέση της ΜΠΕΙ που είναι policy taker και άρα η απάντηση που θα δώσω ε, πρέπει να δίνεται από την Κομισιόν. Άρα πώς να σας απαντήσω. Τέλος πάντων σας ενημερώνω ότι η, η ΜΠΕΙ η ΕΤΕ δηλαδή έχει ως βάση των ενεργειών της το άρθρο 6, δηλαδή λύση με βάση την αγορά. Και κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια γνωμοδότηση όταν ολοκληρωθούν οι εργασίε μας σχετικέ και αυτό θα, θα γίνει με τρόπο πολυμερή. Α, πολύ ενδιαφέρον το πρώτο πάνελ και τώρα για την υπόλοιπη συνάντησή μας. Κύριε Αρτουή, αγαπητέ Πρόεδρε, έχετε τη Ευχαριστώ. Αγαπητή Πρόεδρε, τώρα έχω εγώ την τιμή να παρουσιάσω το δεύτερο πάνελ. Το δεύτερο πάνελ, το οποίο ονομάζεται «Η ένταξη του κλίματος στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020» σε σχέση με τα θέματα τα κλιματικά. Οριζόντιες προτεραιότητες το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 2020-2027 και τώρα ευθύς αμέσως τον λόγο έχει ο πρώτος μας προσκεκλημένος ο Γιώχαν Ορέιλ που ασκεί καθήκοντα διευθύντου στην Γενική Διεύθυνση για τα Δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στο πάνελ για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης για τα δημοσιονομικά. Έχω εδώ κάποιες διαφάνειες, ούτω ώστε να πλαισιώσουν την σύντομη παρέμβασή μου. Α, το ήδη λειτουργεί η οθόνη, πολύ καλό αυτό. Ο συνάδελφος από τα κλιματολογικά, ο κύριος Σόβεν, εστιάστηκε στην πολιτική και στις πολιτικές προτεραιότητες, οπότε εγώ θα περιοριστώ στα θέματα δημιουργικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την ένταξη του κλίματος στις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει τη δράση και το κλίμα μέχρι του 20% του συνόλου του πολίτους πλασίου. Και αυτό το φιλόδοξο στόχο για να μπορέσουμε το mainstream να το υποστηρίξουμε. Αυτό από πλευρά προπολογισμού σημαίνει ότι ο στόχος μας μεταφράζεται σε λίγο παραπάνω από 200 δις ευρώ από το σύνολο του ενός τρεις που προβλέπονται στο τρέχον πολιτές ε, πλαίσιο για την περίοδο 14-20 όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Και τώρα, για να ρίξουμε μια ματιά στην επιλεγή σας μεθοδολογία πρώτα-πρώτα είναι σημαντικό να αναδείξουμε το ότι τα μέτρα αυτά αφορά τις δραστηριότητε και όχι τις επιδόσεις. Δηλαδή, θέλουμε να προσαρμόσουμε τα κριτήρια του ΩΣΑ από τη σύνδεση του Ρίου και να προσαρμοστεί με τις ιδιωτυπίες που έχει ο κοινωνικό προπολογισμό. Και αυτή είναι η γενικότερη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η κλιματική δείκτες ας πούμε. Και υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ πρωτογενών και σημαντικών όσον αφορά αυτές αυτούς τους δείκτες δαπανών και αντιστοιχούν στο 100 και 40%. Επί του συνόλου των δαπανών σε σχέση με το κλίμα. Και έχουμε μία ποικιλία διαδικασιών υλοποίησης. Όλα αυτά είναι γενή σε μια προσέγγιση στιγμή Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε για το ύψος των δαπανών απόλυτα ακριβείς. Οπότε ό,τι ποσά και να επισημάνουμε με κάποιες μεθοδολογίες για κάποιους συντονιστές των πραγματικών δικτών όλα αυτά είναι σε επίπεδο προσεγγιστικό και όλα αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με επιφύλαξη. Για να δούμε τώρα κάποια αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα σε κάθε πολιετές πλαίσιο. Η την περίοδο 14-17 ξεκινούμε. Το σύνολο της δαπάνης για το κλίμα κατά μεσόρο ήταν το 18% του προϋπολογισμού. Και τα προγνωστικά σήμερα για τα υπόλοιπα τρία χρόνια αυτού του MFF, δηλαδή 18 με 20 σημαίνει μια μικρή αύξηση του 18% τα πρώτα 4 χρόνια που θα πάει στο 19,7% για αυτή την τριετία. Ήταν 18, θα πάει 19,7. Όσο κατά αυτό το MFF. Οπότε για το σύνολο ε, του πολιτικού πλαισίου όλη την επταετία, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια ότι το τμήμα αυτών είναι απλά προγνωστικά, οι δαπάνε για το κλίμα όσον αφορά τι πιστό υποχρεώσεων θα μπορούσαν να φτάσει μέχρι το 18,8% του κοινοτικού προπολογισμού. Δηλαδή λίγο πιο κάτω από το 19% ενώ αυτό ίσως δεν είναι η τέλεια επίδοση γιατί η φιλοδοξία ήταν το 20% όμως δείχνει ότι όχι μόνο έχουμε σωστή ρότα, αλλά και για το ότι ε, έχουμε θετική εξέλιξη. Και αν δούμε τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες αυτές τις δαπάνες, αν κάνουμε την αναζήτηση είπε ένα πρόγραμμα και συμπαθάτε με για όλα αυτά τα νούμερα στη διαφάνεια, αλλά από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ήξερα, ε, οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή θέλανε λεπτομερείς ε, πληροφορίες αναταμείο και έτος ούτως ώστε αυτά να τα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Άρα, αναταμείο, το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά το 1β, 2 και το 1α ως κεφάλαιο του πλαισίου. Και οι βασικοί συντελεστές των ε, δαπανών έχουν να κάνουν με το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης που πάει στο 28% του συνόλου των δαπανών που έχουμε ψημένει Επίσης, 23% το EAGF και το 1Β είναι τα διευθυντικά ταμεία για την συνοχή, ενώ το Ταμείο Ανάπτυξης της ε, ε, περιφέρεια 18% και 9% ταμείο συνοχή. Και στο κεφάλαιο 1α κατεβαίνουμε λίγο στα ποσοστά, αλλά πάλι είναι σημαντικά τα ποσά. Το Horizon 2020 έδωσε το 8% του συνόλου και το πρόγραμμα Connecting Europe 6%. Τέλος, η δάλα κεφάλι του πολιτού πλαισίου συνέβαλαν κατά 7,2%. Οπότε κεφάλαια 2, 1β και 1α ήταν το 90% και άνω των δαπανών για το κλίμα. Στο σύνολο δε, ιδίω το δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή ανάπτυξη της ε, υπέδρου και ταμείο γεωργικών εγγύσεων ήταν το 50% του συνόλου. Αυτό σημαίνει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πολιτές πλαίσιο, το όπως τα είπε και ο κύριος Σόβεν και το live εδώ, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα είχε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και τώρα, να στραφούμε σε κάποια σύντομη αξιολόγηση. αφορά τη μεθοδολογία, όσον αφορά το που προσπάσαμε, γιατί γενικώ θεωρεί η Κομισιόν ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και οι εξωτερικοί σύμβουλοι μας είπαν μπράβο για την μεθοδολογία και για την ιστορική συνέπεια αυτού του συστήματος κατανομής των δαπανών για το κλίμα και θέλουμε να δώσουμε κίνητρα όσον αφορά ε, το πόσο το κλίμα θα μπει στις πολιτικές στη φάση του προγραμματισμού. Ε, το πετύχαμε αυτό. Είναι σαφές. Άρα είμαστε σε σωστό δρόμο. Αν κάτσουμε τώρα και συγκρίνουμε το σχεδόν 19% που προσδοκάται να πετύχουμε με αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο και το συγκρίνουμε την περίοδο 7-13, εκεί που είχαμε μέσο όρο μόνο 7%, βλέπουμε ότι υπερδιπλασιάσαμε την επίδοση σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα δούμε τι μαθήματα, τι συμπεράσματα αντιλήσαμε. Αυτό που ειχαμε μεσα ορο μονο 7 βλεπουμε οτι υπερδιπλασιασαμε την επιδοση σε αυτο το δημοσιονομικο πλαισιο τωρα δουμε τι μαθηματα τι συμπερασματα αντιλησαμε αυτο που εξης να αναφέρουμε είναι ότι ο στόχος του ορίζοντα 2020 του 35% δεν επετεύχθη και για το τρέχον πολίτες πλαίσιο περιμένουμε το ράζουν να κινηθεί στο 30 έως 31% των δαπανών για το κλίμα. Αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει προβλεψιμότητα για τα διάφορα στοιχεία του προγράμματος, άρα θα μας προβληματίσει για το μέλλον πώς οι στόχοι για το κλίμα θα πρέπει πλέον να μην εστιάζονται, να μην υποστηριζόνται προς αντίστοιχα τμήματα προγραμμάτων. Το live θα μπορούσε να παίξει πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον, να συμβάλλει περισσότερο στο mainstreaming της υπόθεσης κλιματική αλλαγή. Τώρα όσον αφορά τη μεθολογία της Κομισιόν, είναι τέλεια ε, όχι, βέβαια, τίποτα δεν είναι και όλα επιδέχονται επικρίσεις. Όλα επιδέχονται βελτιώσεις, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή της τωρινής μεθοδολογίας της Κομισιόν θεωρώ ότι προϋποθέτει μία σφαιρική, μία γενική αξιολόγηση. Και οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί επί τη βάση του τι είδους γραφειοκρατία μπορεί να γεννηθεί γιατί υπάρχει συνένεση από όλους μας ότι χρειάζεται απλούστευση. Να μην το ξεχνούμε αυτό και εν κατακλείδη νομίζω ότι τελικά η επιτυχία ή η αποτυχία της υπόθεσης mainstreaming μπορεί να εξεταστεί μόνο με περισσότερα στοιχεία και σε περισσότερο βάθος χρόνου. Ήδη στην προηγούμενη ζήτηση του πάνελ είπαμε επανειλημμένα ότι τώρα μελετούμε την πρόταση για το νέο δημοσιογραφικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί στις 2 Μαΐου. Ε, βέβαια και από τώρα δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες, ούτε μπορώ να περιγράψω και να κάνω προγνωστικά για τα επιμέρους κομμάτια τι θα γίνει και με, τις, με τους ιδίους πόρους. Πάντως το μήνυμα του Κοινοβουλίου αφορούσε το πόσο σημαντική είναι αυτή η νέη ήδη πόρη. Ε, αυτό το αφουγκραστήκαμε, αυτό το καταλάβαμε στην Κομισιόν και το λάβαμε υπόψη στα σοβαρά όταν συνθέσαμε τις προτάσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρέλ. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι στο επόμενο πολιετές θα υπάρχει ένα ξεχωριστός τίτλος κλίμα, μοναδικός. Ε, μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε σε αυτή την ερώτηση αργότερα. Προηγουμένως θα δώσω το λόγο στον κύριο Όουεν, που είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και έρχεται από το Λουξεμβούργο και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Thank you, Chair, for this opportunity to share our work and σας ευχαριστώ Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας και τις εργασίες μας. Έχω και εγώ διαφάνειες. Θα αναφερθώ πρώτα στην έκθεση του Νοεμβρίου 2016 ε, το 20% των πόρων αφιερώθηκαν στην κλιματική αλλαγή. Μετά θα μιλήσω για ε, τη δημοσίευση του 2017 του Σεπτεμβρίου ε, σχετικά. Ε, πρώτον, one in five λέγεται. Βασική ερώτηση. Ο στόχος του 20% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι πιθανό να καλυφθεί για την κλιματική αλλαγή και υπάρχει προστιθέμενη αξία από την προσέγγιση. 200 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν σε όλη την περίοδο για την ναι, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι ε, το Φεβρουάριο του 2016 πήγαμε στην Πολωνία με θέμα τη συνοχή και την ΚΑΠ, στη Γερμανία, Ρουμανία συνοχή και στη Γαλλία, Ισπανία για την κοινή γεωργική πολιτική. Αντίστοιχα ε, είχαμε ελεγκτικό έργο για το ορίζοντα 2020, την Αλία, το πρόγραμμα LIFE και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω συναντηθεί με βασικούς επιτρόπους. Δεν εξετάσαμε ε, τις αρνητικές επιπτώσεις κάποιων δαπανών για την κλιματική αλλαγή ή θέματα ε, του προπολογισμού που δεν είχαν σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Και αντίστοιχα δεν εξετάσαμε άλλη κλιματική χρηματοδότηση εκτός της Ευρωπαϊκής ε, χρηματοδότηση, ας πούμε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής μας. Και δεν καλύψαμε και τις τρέχουσες δαπάνες, γιατί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει προγραμματισμένες δαπάνες και στο πλαίσιο του ε, παρόντος PDP ε, ήμασταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Τι διαπιστώσαμε, ότι είναι το έργο αυτό φιλόδοξο, ότι έχει γίνει πρόοδος, έχουμε περισσότερη δράση, πιο στοχευμένη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιβαλλοντικής, ε, Περιφερειακής Συγγνώμη, Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής. Αλλά στην Γεωργία Ανάπτυξη Πέθρου Αλία και το ΕΚΤ δεν ε, είδαμε σημαντική μετατόπιση υπέρ της κλιματικής δράσης, ούτε να αξιοποιείται πλήρως όλο το δυναμικό και η ε, έρευνα υπολείπεται κατά πολύ του στόχου του 35% όπως ακούσαμε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε ε, ο προϋπολογισμός αυτός στην ε, τρέχουσα περίοδο και ξεπέρασε το 20% το 2016 ήταν πάνω από 20%. Ωστόσο η κατάσταση προβλέψεων για το 2017 και το 2018 και οι υπολογισμοί είναι κάτω του 20% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνολικά εκτιμά ότι αν δούμε ολόκληρη την επταετή προγραμματική περίοδο είμαστε στο 18,8%. 11 με 12 δις δηλαδή λοιπόν από το στόχο που είχαμε. Ε, Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτά τα στοιχεία και στην έκθεσή μας θεωρούμε ότι είναι και υπερεκτιμημένα. Θα σας εξηγήσω. Θα αναλύσαμε τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπαμε ότι δεν θεωρούμε ότι ακολούθησε τη διεθνή ε, καθοδήγηση. Ιδιαίτερα στη γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου ε, έχουν υπολογίσει 33 δις λιγότερο για την περίοδο αυτή. Αυτό αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και δεν ε, εξηγείται επαρκώς εάν ε, δούμε ε, ότι ισχύει εδώ η αρχή της συντηρητικής δαπάνης. Και στην ανάπτυξη της υπαίθρου είδαμε ότι υπάρχουν υπερεκτιμήσεις της τάξης του 24. 24 δι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί μεθοδολογία που δεν κάνει διακρίσεις σαφείς ανάμεσα στα διάφορα μέτρα. Το ίδιο είδαμε και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής. Άλλο τμήμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής κατάφερε, χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία, να ακολουθήσει ε, διαφορετική μέθοδο. Ακόμα έχουμε χρόνο για να γίνουν αλλαγές και στο τρέχον PDP ε, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα μπορούσε αυτό να το κάνει ε, με νέους στόχους ή με αναδιάταξη των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρόν της έργο για ε, το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής για να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες εκθέσεις, η ε, ειδική έκθεση που έχουμε για το προσύνισμα της ΚΑΠ και το σχήμα βασικών πληρωμών του περασμένου Δεκεμβρίου και του φετινού Μαρτίου. Έχουμε έγγραφο ενημέρωσης για τη χρηματοδότηση ε, της Ένωσης του Φεβρουαρίου του 2018 και η χρηματοδότηση και πάλι της ε, μελλοντικής ΚΑΠ. Ορίζον 2020 υπολείπονται κατά πολύ του στόχου του 20% και θα χρειάζεται η μισή τουλάχιστον έρευνα να αφιερωθεί στο κλίμα ε, το επόμενο διάστημα για να ε, καλύψει το κενό. Συστάσεις. Είπαμε ότι είναι καλή αρχή, αλλά χωράει βελτίωση για το μέλλον. Οι συστάσεις 1 και 2 έχουν να κάνουν με τη βελτίωση ε, του τρόπου αναφοράς και των εκθέσεων. Η τρίτη σύσταση λέει ότι θα πρέπει Κατά το σχεδιασμό κάθε γραμμή του προπολογισμού θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασίζεται ε, σε γερή εκτίμηση των αναγκών ανάλογα με την κλιματική αλλαγή και το πώς μπορεί η κάθε περιοχή να συμβάλλει. Τέταρτη σύσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να διορθώσουν τις υπερεκτιμήσεις στην ανάπτυξη πέθρου. Σύσταση πέμπτη, κάθε φορά που βλέπουμε ότι δεν συμφωνεί ο στόχος με το αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί ένα σχέδιο δράσης για να μας πει πώς θα βεβαιωθεί ότι θα καλύψει το κενό και τα ελλείμματα. Ε, Έκτη σύσταση. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, σε διαχείριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα αναλογικό και εναρμονισμένο ε, για έλεγχο της υλοποίησης κλιματικής δράσης. Και μαζί με έναν προεπολογισμό στοχευμένο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα να ε, υπάρξει πραγματική μετατόπιση για την καταπολέμηση κλιματικής ε, αλλαγής, ας πούμε για τη μείωση των ε, εκπομπών αερίου, θερμοκηπίου. Αυτό έχει να κάνει ε, με τον προϋπολογισμό βάση επιδόσεων. Και βεβαίως να διευκολύνεται η μετατόπιση και η ανταλλαγή των καλών πρακτικών. Επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίζει τους τομείς που έχουν υπόαπορρόφηση ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αναπτύξει σχέδια δράσης για να αυξηθεί η συνεισφορά τους. Οι ε, Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν ε, στη γεωργία, ε, στην ανάπτυξη πέθρου και στην αλία της προσπάθειές τους. Ας πούμε, με την εκπόνηση νέων μέτρων ή την αναδιάταξη παλαιών. Εμείς ως ελεγκτές είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κίνδυνος να μην καλυφθεί ο στόχος του 1 στα 5 το 20% μπορεί να έχει γίνει κάποια πρόοδος, αλλά σε τομείς ε, βασικούς χρηματοδότησης δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Θα πρέπει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες και να βεβαιωθούν ότι θα μετατοπιστεί η χρηματοδότηση προς την ε, κλιματική δράση. Γενικότερα κάναμε μια πρόσφατη έρευνα για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή το Σεπτέμβριο, μια γενική επισκόπηση ε, όλης της ελεκτικής που είχαμε κάνει την τελευταία πέντα ετία, όχι μόνο εμείς αλλά και εθνικές ε, αρχές λογιστικού ελέγχου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το μέλλον, τι δείχνει αυτή η γραφική παράσταση, ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο στην καταπολέμηση των αερίων του θερμοκηπίου για τους στόχους του 2020 και του 2030, 20 και 40% αντίστοιχα. Και μέχρι το 2050 η πρόθεση είναι να έχει βιωθεί αυτό κατά 80 με 90% με σημείο αναφοράς στις τιμές του 1990. 1% το χρόνο έχουμε καταφέρει να μειώσουμε ε, τα αέρια της θερμοκηπίου στην πρώτη δεκαπενταετία του 2000, 2015. Μάλλον, μέχρι το 2015 ήταν 1% η μείωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει 1,5% και μέχρι το 2030 τριπλάσια με τετραπλάσια μείωση. Ε, του μέσου όρου για να φτάσουμε στους στόχους του 2050. Αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει τους στόχους εάν δεν κάνει σημαντικές επιπρόσθετες προσπάθειες και αυτό σημαίνει ριζικές αλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και μεγαλύτερη εστίαση στο τι μπορεί να κάνει ε, ο προπολογισμό και ο κρατικός και ε, ο ιδιωτικός και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ τις δύο επιτροπές σας για τη σημερινή συζήτηση. Τελευταία διαφάνεια. Θα πρέπει να δούμε και τη δυσκολία της χρηματοδότησης και το πρόβλημα αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έχουμε εντοπίσει εμείς 7 δυσκολίες ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί και το Κοινοβούλιο. Βλέπετε η χρηματοδότηση είναι ένα από τα επτά προβλήματα, ας πούμε. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται ε, αποκομμένο και απομονωμένο από τα τα, τα συνολικά τα έξι υπόλοιπα, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα αυτά. Ας πούμε, για εσάς τους νομοθέτες είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο ε, στα πλαίσια της σημερινής σας δράση στο λεγόμενο ε, χειμερινό πακέτο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, για την ενεργειακή μετάβαση. Θα πρέπει ιδιαίτερα να ε, είναι τα κίνητρα τέτοια έτσι ώστε να ε, προσελκύσουν ιδιωτικέ επενδύσει πολύ περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε λοιπόν. Κάνατε έναν έλεγχο και επί κάποιων σημείων υπάρχει κάποια διακοσμητική προσέγγιση αν θέλετε, κάλυψης. Ευχάριστη παρουσίαση. Αλλά φαίνεται σαν λίγο ότι έχει υποστεί κάποια... Είναι κάπως θεσιδωμένη παρουσίαση. Ο κ. Μάκος Ρίλινγκ, συντονιστής Finance και επιδοτήσεων, ο κ. Μάρκος Τρίλινγκ του Climate Action Network. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω κάποιες λεπτομέρειες. Να διαβάσετε μέσα από τις γραμμές. Κυρίως βλέπουμε πόσο είδαμε κάποια αυτιασυδωμένα στοιχεία Έχουμε 150 ομάδες εμείς ε, σε όλη την Ευρώπη, στο Climate Action Network. Ποια είναι η αποστολή μας? Να εμποδίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα, επικίνδυνα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος. Εξετάσαμε διάφορα προγράμματα, το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, και εντοπίσαμε δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται, δυνατότητες, πώς ο προπολογισμό μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις αλλαγές του κλίματος, ε, συναγάγαμε κάποια συμπεράσματα, πήραμε μαθήματα, αυτά μεταφράστηκαν σε ένα όραμα για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό θα σας παρουσιάσω. Καταρχάς, ο λόγος ε, παρουσίας μας εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι η Συμφωνία των Παρισίων, άρθρο 2 και τι απαιτεί οικονομικές ροές ε, που πρέπει να διατίθεται για να σταματήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Και είναι τεράστια οικονομική ροή προβλησμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεις. Κάθε κονδύλι, κάθε α, ε, δαπάνη πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο συνάδει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Αυτή είναι η θέση μας. Ο συνάδελφος του Ελεκτικού Συνεδρίου έδειξε ήδη φωτογράφημα Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να μειώσουμε και με δραματικό τρόπο τι ανθρωπογόνες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για να πετύχουμε το στόχο του 20% ε, αναφέρθηκε ότι ο στόχο του 40% δεν θα καλυφθεί με, την, με τον παρόντα αριθμό μειώσεως. Και ξέρουμε ότι πολύ μεγαλύτερε προσπάθειες απαιτούνται για να πετύχουμε την μείωση 80 με 95%. Τι θα σας δείξω τώρα. Ότι αυτές οι επιταχυμένες προσπάθειες που απαιτούνται μπορούν να γίνουν με την βοήθεια του προπολογισμού. Και ένας ο υπολογισμό με βάση το κλίμα μπορεί να κάνει τη μετάβαση πιο ομαλή και να δώσει όθηση, κατάλληλη όθηση που απαιτείται για να περικοπούν οι εκπομπές αρήνου θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι κατά τομέα εκπομπές αρήνου θερμοκηπίου στην Ευρώπη το έτος 2015. Αυτό αντιμετωπίζουμε και όπως σας ε, δείχνω, είναι επιλέξιμη η τομή για χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για κάποιους τομείς, η χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, είναι αποφασιστικός παράγων για την ε, ύπαρξη ή καταστροφή ενός τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει για την πολιτική συνοχή πρόταση αρχές Μαΐου, αλλά προπολογισμό βεβαίως αποτελείται από το άθροισμα των προγραμμάτων του και πιστεύουμε και περιμένουμε η πολιτική συνοχής που θα δοθεί τον ε, μήνα Μάιο και στον προγραμματισμό ότι θα ληφθεί κατάλληλη απόφαση. Κατά πόσο χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής ε, δίνεται για αποτέφρωση αποβλήτων ή για ε, ανακύκλωση, για την κυκλική οικονομία. Η πολιτική συνοχής, η χρηματοδότησή της τώρα στις χώρες συνοχής κυρίως χρηματοδοτεί υποδομές οδικές, το μεταφορικό τομέα. Αν θέλουμε να μειώσουμε την αύξηση των εκπομπών των μεταφορών, πρέπει να αποφασίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιοι θα είναι οι όροι για μελλοντική χρηματοδότηση. Βασικές υποδομές ή μέτρα που προωθούν βιώσιμη κινητικότητα για αγαθά και ανθρώπους και μετάβαση προς αυτό το στόχο. Η πολιτική συνοχής επενδύει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Κτίρια πρέπει να μειώσουν, έχουμε το 12% πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές των αερίου θερμοκηπίου. Στις οικοδομές υπάρχει μεγάλη δυνατότητα στα κτίρια να πετύχουμε στόχους μέσω χρηματοδοτήσεως. Άλλο παράδειγμα, το μέσο για τη της Ευρώπης, Connecting Europe Facility. βλέπουμε να κινούμεθα περισσότερο προς το φυσικό αέριο. Χρηματοδοτείται δύο φορές παραπάνω το φυσικό αέριο εν συγκρίση με την ηλεκτροδότηση. Ξέρουμε ότι συμφορήσει στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι ότι χρησιμοποιούμε Δεν βάζουμε ε, την ενέργεια που παράγεται από ανεμοστρόβιλους ή από, τα, από τους ηλιακούς ισορρευτές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα μειώνει εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου και αερίων που δεν ανήκουν στα αερία του θερμοκηπίου. Έρευνα και καινοτομία. Για πρώτη φορά αυξάνονται οι εκπομπές ε, του, ε, των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα του ETS. Αν θέλουμε να ηγηθεί βιομηχανικά η Ευρώπη μέσω καθαρών τεχνολογιών και κάνοντας σωστή μετάβαση, τότε χρειάζεται έρευνα και καινοτομία και τα σχετικά προγράμματα. Πολιτική συνοχής, επενδυτικό εργαλείο για τους τομείς που εμπίπτουν στην απόφαση για επιμερισμό των προσπαθειών. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες η πολιτική συνοχή και η σχετική χρηματοδότηση είναι το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης δημοσίων υποδομών. Βλέπετε τα διαθωτικά ταμεία, το ποσοστό διαθωτικών ταμείων στις δαπάνες, πώς συμμετέχουν. 12 χώρες, ε, σε 12 χώρες πάνε μέχρι 40% χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εικόνα έχουμε το πλαίσιο που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη δανειοδότηση, που ε, επηρεάζει την ιδιωτική επένδυση. Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε αυτές τις περιοχές επηρεάζει και το πώς θα αναπτυχθούν οικονομικά οι περιοχές. Μέσω όρο των χωρών βλέπουμε εδώ πώς κατανέμονται οι πόροι από το Ταμείο Συνοχής. Στήριξη επιχειρήσεων, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε κοινωνική ένταξη, κατάρτιση, απασχόληση, μεταφορές 20% βλέπετε, περιβάλλον 10%, ενέργεια 8% κλπ. Από κοντά αν κοιτάξουν τα στοιχεία. Τη δαπάνες 8% για την ενέργεια. Βλέπουμε φυσικό αέριο, ε, έχουμε ακόμα χρησιμοποιούμε ρηχτά καύσιμα. Το μεγαλύτερο κομμάτι των δαπανών για την ενέργεια πάει στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμως, στην απόδοση των κτηρίων. Περίπου 4% της χρηματοδοτήσεως συνοχής δαπανάται στα κτίρια. Έχουμε πολλές δυνατότητες εκεί. Μετά, βλέποντας τι γίνεται με τη μετάβαση στον αφορά το υλικό που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευφυής διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στην πολιτική συνοχής. 5,4% είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης. Δεν ότι δεν πάνε τα περισσότερα χρήματα στην ε, μετάβαση προς καθαρή ενέργεια, στις μεταφορές. 20% της πολιτικής συνοχής με ένα σχόλιο όπου οι οδικές κατασκευές, οι αυτοκινητόδρομοι δεν καλύπτονται. Το μεγαλύτερο κομμάτι των μεταφορικών υποδομών πάει στο σιδηρόδρομο και στι οδικές μεταφορές. Το ερώτημα είναι όμως η χρηματοδότηση για τη μετάβαση που πάει στο μεταφορικό τομέα, για λύσεις κινητικότητας που συμπεριλαμβάνουν την αστική διάσταση που θα πρέπει να εξετάζει και τη μεταφορά των αγαθών. Εδώ έχουμε το μέσο για διασύνδεση της Ευρώπης. Μεταφορές. Χρηματοδοτούμε σιδηροδρόμους κυρίως και έχουμε δύο φορές παραπάνω αγωγούς φυσικού αερίου από τη διασύνδεση ηλεκτρική. Ενώ προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τη διασύνδεση. Επιδοτήσει για το ρηχτά καύσιμα δεν ταιριάζουν συμφωνία των Παρισίων. Έχουμε υποστήριξη για υποδομέ για φυσικό αέριο σε πολλά προγράμματα με 200 δι. Επιταχύνω, επιταχύνω. 20% δράση για το κλίμα, τα ακούσαμε αυτό, 106 δισεκατομμύρια στην κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλουμε να ακολουθούμε δράση για το κλίμα που κάνει την αλλαγή, βελτιώνει. Τα υπόλοιπα 40 δις από ε, υποδομές υδρομικές. Πολύ σημαντικό. Όταν εξετάζουμε τον εξοπλισμό για τη μετάβαση όσον αφορά την κινητικότητα και όσον αφορά την ενέργεια, μπορούμε να βελτιώσουμε την χρηματοδότηση, να αυξήσουμε. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική δράση για το κλίμα. Να αφήσουμε εκτός τι υποδομέ το φυσικό αέριο και υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σε βασικούς τομείς να λάβουμε δράση για το κλίμα και σε βασικέ περιοχέ. Πώ θα τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε υψηλότερους στόχους για προχρηματοδότηση, για προσημείωση ποσών για το κλίμα. Το συζητήσαμε. Να βελτιώσουμε λοιπόν τις επιδόσεις των προγραμμάτων το κλίμα, να αυξήσουμε το χρήμα που θα δώσουμε για ευφυή ε, διανομή του ηλεκτρικού ρεύματο και διάφορα άλλα μέτρα και θα πρέπει να έχουμε μεθοδολογία να ελέγχουμε κατά πόσο χρησιμοποιούμε σωστά τα προγράμματα για την μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και θα πρέπει όσο ο να τα λαμβάνει αυτά υπόψη να λαμβάνει υπόψη το κλίμα. Να μην χρηματοδοτούμε φέρον το φυσικό αέριο, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ και να ευθυγραμμίσουμε τι μεταφορέ και τι επενδύσει με τη μείωση εκπομπών του αερίου, του θερμοκηπίου με κατάλληλα προγράμματα ηλεκτροδότηση και στρατηγικέ για μείωση τη χρήση ε, ορυκτών καυσίμων. Τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό. Οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω πρέπει να ταιριάζουν με, με αυτά που δαπανούν τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε μακροπρόθεσμα συστηματικά την προσέγγιση. Και επόμενη ευκαιρία θα είναι τα σχέδια για το 2030 τεχνικά. Και θα πρέπει εκεί να δούμε τι δεσμές θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη για την επιτυχία των στόχων τους. Αποθεματικό για επιδόσεις, μηχανισμοί που δίνουν κίνητρα πρέπει να εφαρμοστούν, να αυξηθούν οι φιλοδοξίες. Κλείνοντας, ο προϋπολογισμός είναι μικρό σε συγκρίση με άλλε οικονομικέ ροέ, είναι όμω σημαντικό για βασικού τομεί όπω η γεωργία, οι μεταφορέ, η ενέργεια, η ζωή στα πόλει και σε, σε περιοχές αποδέκτες, κυρίως λιγότερο ανεπτυγμένε περιφέρειες, στα ανατολικά. Ε, υπάρχει δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται, σημαντικό, για να αυξήσουμε τις δράσεις για το κλίμα και δεν πρέπει να κάνουμε επανάσταση, μπορούμε να βασιστούμε στις υφιστάμενες υποδομές στις προσημειώσεις ποσών, κίνητρα που θα δίνονται, ρεσιμότητα και πολύ σημαντικό, στατηγικός και επιχειρησιακός, ε, ε, στατηγική και επιχειρησιακή διασύνδεση με τα προγράμματα τα εθνικά για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το όραμα αυτό που παρουσιάσατε. Πολύ αισιόδοξο. Μας αφήνει σημαντικά περιθώρια για πρόοδο. Καλώς. Πάμε σε ερωτήσεις. Όποιος επιθυμεί να αντιδράσει σε αυτά που παρουσιάστηκαν, στις τρεις παρουσιάσεις, που ήταν άκρως διαφωτιστικές. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον κάθε ε, καλεσμένο μου φαρενεύει. Ο πρώτος παρακαλώ. Okay, um, several things come Αναδύονται διάφορα ζητήματα, λέει ο κ. Πρώτα πρώτα. Διάβασα με ναι, ενδιαφέρον την έκθεση του ελληνικού συνεδρίου. Α, και όταν μιλήσαμε για το μέλλον των ειδών διατροφή, για το πρασίνισμα τη ΚΑΠ, την αποτελεσματικότητα, είχαμε αφήσει το κείμενο σήμερα το πρωί για την πράσινη χρηματοδότηση. Αυτό μου θα τώρα το μυαλό. και άμα τη διαβάσει κανείς ε, προσεκτικά, καταλαβεί ότι τελικά μόνο όνομα κάνουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Τις βάζουμε την ετικέτα απλώς. Δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν γίνεται ο μετασχηματισμός που επίδει ακόμα. Δεν ξέρω, το κατάλαβα καλά. Αν όχι, μάλλον αν το κατάλαβα καλά, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε. Κατά δεύτερο λόγο, όσον αφορά το πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της χρηματοδότησης για μια αλλαγή στην πολιτική μεταφορών και στα δίκτυα, ισχύει ή όχι. θέλουμε να πετύχουμε επιπτώσεις για πρασίνισμα και έτσι να έχουμε νέους μηχανισμούς κατανομής οπότε να φτάσουμε σε αποτελεσματική χρήση κάποιων οχημάτων όπως τα ηλεκτρικά αλλιώς εναλλακτικά τι πώς αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν αποτελεσματικά τα δίκτυα σε σχέση με τον υπολογισμό. και για την πολιτική συνοχή. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιο προγράμματα και έργα ε, χωρίς να χρησιμοποιούμε ε, υδρογονάνθρακες. Επίσης, λέμε, ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε αυτό ή εκείνο το ποσό να είναι διαθέσιμο στο πολιτέ πλαίσιο, στον προπολογισμό ως ποσοστό, ούτω ώστε να πάνε αυτά τα λεφτά για την αλλαγή του κλίματος. Όμως, το αποτέλεσμα της επιδοηλοποίησης μου φαίνεται ότι είναι ανεπαρκές. Εμείς ως νομοθέτες, ως πολιτική, πώς μπορούμε όταν κάνουμε αποτελεσματικά να διαρθρώσουμε εκ νέου τον ε, προϋπολογισμό, να βάλουμε καινούργιες αιρεσιμότητες ή ε, εναλλακτικά τι κόλπο μπορούμε να μετέλθουμε τόσο ώστε όλες οι αυτές οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν. La parole est maintenant à la présidente ε, Τώρα η πρόεδρος Γκρέσλε έχει το λόγο. Τα γερμανικά. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αν δούμε τα κτίρια, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και τη χρηματοδότηση μέτρων. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχετε βγάλει εσείς. Γιατί μέχρι τώρα κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Και για τη χρηματοδότηση της ε, καταπολέμησης χρηματικής αλλαγής κάνουμε πολύ μικρά βήματα και απατηλά για το πρασίνισμα υπήρξε ολέθρια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω. Γιατί κάνουμε πολύ φασαρία. Και μεγάλα λόγια λέμε, σε καμία περίπτωση αυτά όμως δεν ε, συμπίπτουν με τα έργα. Άλλος κανείς, ο κύριος Τάραντ. Yeah, I have... Um, Πολύ σύντομα έχω δύο ερωτήσει για την Επιτροπή. Μία γενικής υφή Συμφωνεί με αυτό που είπε το Ελληνικό συνέδριο ότι απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Συμφωνείτε ναι ή όχι. Επίσης, για αυτό το πρόγραμμα, το live, τι προοπτικέ έχει για το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και μια σύντομη για το Ελληνικό συνέδριο. Έχετε συστήσει ποτέ ότι θα πρέπει να υπάρχει οικονομικό έλεγχο για το τμήμα του προπολογισμού που είναι άσχετο με το κλίμα. Γιατί και αυτό θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα όσον αφορά τι προσπάθειε για την αλλαγή του κλίματο. Καμία ερώτηση προ τον κύριο Τρίλινγκ. Γιατί Ευχαριστώ για τον τρόπο που μιλήσατε, γιατί αγγίξατε την οικολογική μου συνείδηση κόντρα σε κάθε πνεύμα πολιτικού συμβιβασμού. Και τώρα, αφού δεν έχει άλλος ερώτηση, να ρωτήσω υποφαινόμενος πρώτα-πρώτα. Με εντυπωσιάζει το ότι θεωρεί η Επιτροπή ότι βρισκόμαστε στο 20% του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οπότε 20% του 1% που είναι 0,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Όμως η επιδόνηση του κλίματος είναι τέτοια που αυτό θα μπορούσε να καταλήξει στο να εξαλειφθεί η ζωή από τον πλανήτη. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα χωρίς προηγούμενο. Είναι το τέλος της ανθρωπότητας, της εξέλιξης. 0,2% του ΑΕΠ για μία προτεραιότητα είναι φραγκοδίφραγκα. Υπάρχουν τα μέτρα, τα μέσα. Μας εξήγησε το ελεγκτικό συνέδριο ότι αυτά είναι κάπως διακοσμητικά, καλοπιστικά. όλα αυτά τα μικροφτιασίδια. Με αυτά θα μπορούσαμε να πάμε στο 0,1-0,15% να κατέβουμε. Μπορούμε στην Ευρώπη να εκμεταλλευτούμε τις προσπάθειες των κρατών μελών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι μετρήσιμο. Μπορείτε να το μετρήσετε. Οπότε τώρα το κοιτάζετε δεν έχουν οι τρεις προσκεκλημένοι μας. Δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτα το λόγο. Εσείς κύριε Γιουρέλ για να, να, να, να, απαντήσετε στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των υπολογισμών σας. Όχι, όχι, δεν τολμώ να κοντράρω το ελληνικό συνέδριο. Λέω κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω πάντως να σας δώσω τρία σημεία. Κάποιοι βουλευτές ερώτησαν το κατά πόσον έχουμε κάτι πετύχει, πώς είναι η κατάσταση. Ε, αυτό εκφεύγει τον χειρό. μου. Εγώ θα σας πω απλώς τι γίνεται με τις δαπάνες για το κλίμα, πώς είναι η κατάσταση. Απλώς μετρούμε την ε, συνεισφορά του προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα δεν το μετρούμε. Άρα τι να πούμε. Τουλάχιστον με αυτόν τον μηχανισμό της παρακολούθησης υποπτήρια, το tracking. Οπότε πάμε στο δεύτερο σημείο. Ε, αν συμφωνούμε με τις επικρίσεις του συνεδρίου. Γνωρίζουμε τις ε, συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου που διατυπώνται στην έκθεση του 16 και θα έχουμε πει διαμακρών με το συνεδρίο και κάποιες από αυτές τις ε, συστάσεις έχουν γίνει αποδεκτές ενώ λόγια Αλλά αφαιρεπήν έχουμε αυτή τη σύσπιση όσον αφορά ε, την, δίθυνη, την ε, πιθανή υπερεκτίμηση όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Παραδεχτήκαμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε κάπως να χτενίσουμε την μεθοδολογία μας από το 21 και μετά. Αλλά δεν βλέπουμε ότι η αλλαγή της μεθοδολογίας θα αποδώσει τώρα ενώ είναι εξελίξει το πολιτές πλαίσιο που θέλουμε να υπάρχει συνέπεια, να υπάρχει ε, διαδοχή ομαλής, στις αξιολογήσεις. Έτσι τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Τώρα, ε, άλλες συστάσεις του συνεδρίου δεν έγινε αποδεκτό, γιατί θεωρήσαμε ότι θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και σε εθνικό επίπεδο Αυτά τα σχετικά δεν τα αποδεχόμεθα. Τώρα το τρίτο που θέλω να σας σχολιάσω έχει σχέση με το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Δημοσιονομική Αρχή. Πέρα το συγκεκριμένο θέμα ε, της παρακολούθησης των δαπανών για το κλίμα, η Μεσονομική Αρχή βεβαίως και θα έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα με τη νέα γενιά των κοινωτικών προγραμμάτων. Οπότε και εμείς θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας ε, το Μάιο και το πρώτο μισό του Ιουνίου. Και βεβαίως έτσι θα αναδειχθεί και το ζήτημα του κλίματος. Βέβαια μπορεί να παρέμβει και η νομοθετική αρχή. Παράδειγμα με το να προταθούν κάποιες ρεσιμότητες κλπ. Και εδώ βάζω τελεία πρόεδρε. Αρτή. Ευχαριστώ κύριε Ιουρέλ. Ο ε, κύριος Βιν Όουεν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που απευθύνατε στο ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Χάουαρθ, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας πρώτα. Για την έκθεσή μας σχετικά με το πρασίνισμα, σας ευχαριστώ που την αναφέρετε. Είναι πρόσφατη και ε, αν θέλετε διαβάστε τη, ε, ε, όσοι δεν έχετε, και ε, πραγματικά Αναποκρίνεται σε αυτά που σας είπαμε το 20% για τη γεωργία και το πρασίνισμα. Η έκθεση για το πρασίνισμα λοιπόν τι έλεγε και παραθέτω όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή είναι απίθανο να ενισχύσει ε, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα περιβαλλοντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επιδείξει αρκετή ε, φιλοδοξία ε, ως προς τους στόχους του πρασινίσματος και δεν πρόκειται να αποδώσει σημαντικούς καρπούς αυτό. Υπάρχουν σημαντικές απώλειες και δεν πρόκειται ε, να αλλάξει ε, συνολικά τον τρόπο εκμετάλλευσης ε, των καλλιεργειών παρά μόνο κατά 5% το πρασίνισμα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε ένα πνεύμα διαρκούς βελτίωσης και εξοικονόμησης πόρων. Έτσι θα πρέπει να ενταχθεί και η έκθεση αυτή στο γενικότερο πλαίσιο ε, του mainstreaming της ένταξης των πολιτικών για το κλίμα στο προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα στα δίκτυα των μεταφορών και ε, αυτό που είπατε για τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα και την υποστήριξή τους και τι πρέπει να κλείνει. Ε, με χαρά φαντάζομαι θα ακούσετε ότι αυτό το καιρό ε, εκπονούμε μια ειδική έκθεση για τη στρατηγική και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μιλώ και για τη στατική αποθήκευση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και την κινητή αποθήκευση σε συσσωρευτές ας πούμε, σε αυτοκίνητα ή άλλα ε, κινούμενα μέσα. Ελπίζω του χρόνου τέτοιου καιρό να μπορέσω να έρθω να απαντήσω ε, σε αυτή την ερώτησή σας ε, με μεγαλύτερη πληρότητα. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες που θα τις μελετήσουμε αν είναι πραγματική στρατηγική και αν πιάνουν τόπο τα χρήματα. Για τη συνοχή τώρα, ρωτήσατε για το πεδίο ε, προσημείωση ειδικών ε, ε, γραμμών του προπολογισμού για την απομάκρυνση μας από την εξάρτηση από το διοξίδιο του άνθρακα. Έχω κάνει δύο ειδικέ εκθέσεις σε αυτό και σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας σε τρία κράτη-μέλη. Γιατί κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψουν την πυρηνική ενέργεια και ξέρουμε ότι υπάρχουν περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η τοπική βιομηχανία, η τοπική κοινωνία και απασχολήσει έχει βαριά εξάρτηση είτε από ε, πυρηνικά εργοστάσια είτε από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα ας πούμε. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ε, μπορεί να χρησιμοποιούνται και αυτό συνιστούμε εμείς ευέλικτα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να υποστηριχθεί και η κοινωνική μετάβαση γιατί ε, ε, αναγκαστούν να κάνουν μεγάλες αλλαγές ιδιαίτερα αυτές οι περιφέρειες. και ε, περιμένω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει κανένας μηχανισμός για τη μεγαλύτερη επιβολή. Οι ελεγκτές τείνουν να επανέρχονται και να εξετάζουν ξανά κάποια πράγματα. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, θα επανέλθουμε μετά από πέντε χρόνια να το τσεκάρουμε. Όπω το θέμα αυτό τη εγκατάλειψη των πυρηνικών εργοστασίων. Και να βεβαιωθούμε ότι το mainstreaming θα προχωρήσει την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Αυτό είναι δικό σα θέμα, όχι δικό μα. Αλλά με χαρά θα δούμε να συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν δεν επανέλθει το ελεγκτικό συνέδριο να δει και κατά πόσο οι συστάσει και η μεθοδολογία του έχουν υλοποιηθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό είναι ένα ένα είδος λογοδοσίας, αλλά βέβαια πραγματικά πρέπει να απαιτείται περισσότερη και καλύτερη μεθοδολογία. αιτήσει, εκθέσεις και ε, πρακτικές τήρησης λογαριασμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογιστικές. Γεια σας κυρία Γκρέσλε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Είστε πρόεδρος της σημαντικότερης επιτροπής ε, στο Κοινοβούλιο. Οι ερωτήσεις σας απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τους αφήσω να απαντήσουν εκείνοι. Ε, κύριε Τάραντ, Ρωτήσατε αν ελέγξαμε ε, το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι το κλιματικό σκέλος. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Εμείς ακούμε ε, όλους τους ενδιαφερομένους στο ετήσιο πρόγραμμά μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σας είπα τι δεν καλύψαμε ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ άρχισα να δουλεύω στη συνοχή Πάντα θα πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις για τη συμβατότητα με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Ακούω να γίνεται μέγας λόγος να γίνει 100% φιλικός ο προπολογισμός και συμβατός με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος λογιστικός έλεγχος, αλλά και συναρπαστικός ταυτόχρονα. Δεν θα σας ε, τάξω τίποτα. Ο Πρόεδρος, κύριε Αρτσουή, κάνατε πολλές ερωτήσεις εκεί τα αρχικά σας σχόλια πριν παρουσιάσω την έκθεσή μου ε, γέννησαν κάποια ερωτήματα και θα ήθελα με ευκαιρία να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν κάναμε έλεγχο. Ε, έχουμε προτείνει σε μελλοντική φάση να ελέγχουμε όλα τα όργανα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Δεν λέμε μην προχωρήσετε στο mainstream, αλλά λέμε ότι έχουν γίνει κάποιες ε, πρόοδοι. Οι μεθοδολογίες φυσικά χωράνε βελτίωση, ιδιαίτερα στη Γεωργία οπωσδήποτε και καλό είναι που ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώνει ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις συστάσεις μας για να βελτιωθεί. Αλλά και στην έρευνα και την καινοτομία ισχύει αυτό ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που δεν είχαν στόχους ειδικού για το κλίμα και όταν το ελέγξαμε διαπιστώσαμε 1,4% του συνολικού ποσού πήγαινε με δράσεις για το κλίμα. Είναι πολύ δύσκολο να, να συγκεραστεί αυτό με ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γενικά για τις δαπάνες για το κλίμα, Πρόεδρε, δεν κάνουμε εμείς το λογιστικό έλεγχο στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουν εξαιρετικού οργανισμού στα κράτη-μέλη και η Γαλλία, το ελεγκτικό συνέδριο, το La Cour de Compte, συνεργάζεται μαζί μα. Αλλά δεν προσθέτουμε τις δαπάνε εκεί, δεν κάνουμε εμεί το λογιστικό έλεγχο των κρατών μελών, απλώς κοιτάμε ποια είναι τα βασικά μηνύματα και ποια είναι τα λύματα και είμαστε σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους, σεβόμενοι πάντα πλήρω την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών να κάνουν το λογιστικό έλεγχο στην επικράτειά τους. Εμείς ελέγχουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ευχαριστώ. Βεβαίως, η εθνική κυριαρχία για τους ελέγχους ε, μπορεί να θα δούμε που θα καταλήξει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει ειλικρίνη αν ονόματι της εθνικής κυριαρχίας. Είναι ενδιαφέρον να υπάρξει μια ελάχιστη σύγκληση των εργασιών και των προδιαγραφών που εφαρμόζεται για να διεξάγετε τους ελέγχους σα και να υπάρχει σφαιρικό όραμα για την Ευρώπη όσον αφορά το κλίμα. Αυτό που παρακάμει 10,15% του προπολογισμού του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού μέσω του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού είναι πολύ στο οριακό. Αν παράλληλα τα κράτη επιμένουν σε δράσεις που πηγαίνουν κατά του κλίματος δεν έχει νόημα η όλη προσπάθεια. Παρά τα αυτά αν θα είχα κάποια σύσταση, μια ευχή να εκφράσω, θα ήταν το λεκτικό συνέδριο να μπορεί να συντονίσει και να προσανατολίσει τι εργασίε που διεξάγονται στους εθνικούς, στα εθνικά Ελεκτικά συνέδρια, φροντίζοντα να υπάρχει η ίδια θεμητή προσέγγιση και σωστή αντιμετώπιση παντού. Να προσθέσω κάτι που θα μπορούσε να μα βοηθήσει να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε και την πρότασή σα εάν προχωρήσουμε στα πλαίσια του ενεργειακού πακέτου και σχετική νομοθεσία οι αξιωματούχοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγαν στα πλαίσια τη του κανονισμού τη Ενεργειακή Ένωση, που υπόκειται σε διαπραγματεύσει τριμερούς διαλόγου, το Συμβούλιο πρότεινε σε απάντηση πρώτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να υποβάλουν ολοκληρωμένα σχέδια για την ενέργεια και για το κλίμα για δεκαετή περίοδο 2021 2030 και μπορεί να υποβάλλονται κάθε διετία εκθέσεις προόδου και μπορεί να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προόδο και να αξιολογήσει χρειάζεται σύσταση υπό συγκεκριμένο κάτω μέλος ή πιο γενικές συστάσεις. Αν ενεργειακά σχέδια αποδεικτούν ότι είναι σε εθνικό επίπεδο ποιοτικά, θα μπορούν να συμπεριλάβουν τα στοιχεία των δαπανών του κράτους μέλους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να σε θέση να αθροίσει τα στοιχεία και τότε μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους. Υπάρχουν πολλά εάν σε αυτή την υπόθεση. Ποιο είναι το πλαίσιο όμως. Με την επιφύλαξη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου που είναι περισσότερο στα δικά σας χέρια από τα δικά μου υπάρχουν προτάσεις που διαμορφώνονται ούτω ώστε να υπάρχει μια γενική επισκόπηση που ίσως να επιδιώκεται. Από τη στιγμή που θα ισχύσει αυτό είναι πολύ ευκολότερο οι ελεγκτές να κινηθούν σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως και τα δύο επίπεδα έχουν ρόλο δραματίσουν να δούμε τι γίνεται. Αναφισβήτητα, μ' αρέσει ε, να συμπεριλαμβάνεται η καινοτομία. Αρχικά θα τα πετυχαίνουν όλοι. Χρειάζονται προσαρμογή και να βοηθήσουμε. Μπορεί να προσθέσουν πρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής κάτι σε αυτά που είπα, αλλά εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την παρούσα πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Όεν. Κύριε Τχίλινγκ, θα ήταν καλό αν ήσασταν λακωνικός. Θα είμαι σύντομο. Ο κύριος Όαν απάντησε την ερώτηση όσον αφορά τι υποδομέ ηλεκτρική ενέργειας στην πολιτική συνοχή και τη μετακίνηση στόχους στην οικονομία χαμηλού άνθρακα. Σχόλιο για την πολιτική συνοχή και πώς μπορεί να αλλάξει δομικά το τοπίο. Υπό κοινή διαχείριση πολιτικής συνοχής από τη στιγμή που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη επί συμπράξεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμογή τους και επιλογή, η επιλογή των προγραμμάτων στα χέρια των κρατών μελών. Τι μπορώ να πω εγώ. Ότι η πολιτική συνοχής, συχνάκης, ε, είναι, είναι στήριξη προϋπολογισμού σφαιρική για τις χώρες. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή, σωστός συντονισμός. για τους στόχους του 2030 μέσω εθνικού σχεδιασμού. Αυτό είναι σημαντικό για να γίνει η μετάβαση, η αλλαγή σε αυτούς τους τομείς. Merci. Nous allons en rester là car le temps malheureusement euh, nous, nous... Μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς και πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η ακρόαση το αργότερο στις 17 και 40. Διότι και 30-40 διότι θα πρέπει 17 17-45 να πάμε σε άλλη αίθουσα για να συναντήσουμε τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το τρίτο τμήμα. Εκεί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι όλες οι δαπάνες του, όλοι οι πόροι του, ευρωπαϊκού προλογισμού να οδηγούν σε προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή σύμφωνα με τις κοινέ προτεραιότητες. Και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα χρονικό το 2030. Για να έχουμε τον κύριο Μωρή Σάφερ, πολιτικό σύμβουλο για ενεργειακά θέματα, ΕΚΟΦΙΣ. Κύριο Σάφερ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην ακρόαση. Και ελπίζουμε ότι θα εντοπίσουμε την προβληματική με τις προτάσεις μας, οπότε ίσως και κάποιες από τις διαφάνειες που θα δούμε, ίσως τις έχετε αντικρίζει. Πρόγραμμα από το ECOFIS που είναι μια εταιρεία consulting παροχής συμβουλών. Έχουμε ε, πέντε έδρες στην Ευρώπη και ε, υπαγόμεθα στην Νάδικαν, την Αμερικανική εταιρεία. Έχουμε 600 ειδικού για κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια και ε, στην ε, Έχουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας όσον αφορά παροχή συμβουλών σχέση με το κλίμα, βιώσιμη ενέργεια για όλους επίσης. Για να δούμε τώρα μερικά σημεία. Ε, μιλούμε για τις ανάγκες τις ε, επενδυτικές ε, που αφορούν το πλαίσιο του 2030, πώς μπορούμε να έχουμε προσθεμένη αξία και Έχουμε τον στόχο του ε, mainstream για το κλίμα, να δούμε τα θέματα επίσης ε, της ε, εποπτείας, παρακολούθησης, απολογισμού για τις δαπάνες για το κλίμα, τους δείκτες, το ενεργειακό αποτύπωμα και να δούμε το live άλλα προγράμματα και κατέβουν σε κάποιες ε, συστάσεις όσον αφορά κάποια έργα, προγράμματα που είναι μικρά, αλλά, αλλά σημαντικά. Να, το live και άλλο ένα. Για μια ευφύ ενέργεια στην Ευρώπη το 2030. Τώρα, τονίζουμε ότι θέλουμε να δούμε ποια είναι η αξία στην Ευρώπη και έχουμε τον στόχο του 40% το 2030 για ανανεώσιμε πηγέ συνεργεία. Ε, είπαμε τουλάχιστον 27% ανανεώσιμα και 27% βελτίωση για την αποδοτικότητα. Και το θέμα είναι εάν και εις ποιο βαθμό μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτούς τους ε, στόχους γιατί αυτό επεφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε για 32% και να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη Συμφωνία των Παρισιών. Έχουμε τώρα αυτή την ε, μελέτη της Ρικάρντο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει για το κενό το επενδυτικό όσον αφορά τους στόχους ενώπιση του 2030 και πρόκειται για 178 δις ευρώ ετησίως επιπρόσθετων δαπανών και αυτό ε, μας τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να κατευθύνονται οι πόροι για πράσινα έργα και προγράμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμη γεωργία και επίσης έτσι φαίνεται το πόσο σημαντικός είναι ο προϋπολογισμός αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει. Ο κύριο Σόβεν στην αρχή μας τα είπε. Από μόνο του προπολογισμό δεν μπορεί να καλύψει όλε τι επενδυτικέ ανάγκε, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί έτσι μοχλεύει ιδιωτική χρηματοδότηση αλλά και κρατική κρατών μελών γιατί καταπολεμεί διάφορους φραγμούς στις επενδύσεις. Θα δούμε έχουμε την ε, προσέγγιση της ε, Κομισιόν για το mainstream του κλίματος και επίσης έχουμε και τη λεγόμενη ποσόστοση για το κλίμα που είναι ο ελάχιστος ε, στόχος δαπανών και αυτό είναι κάτι σαν ένα παράδειγμα προς για τα κράτη-μέλη σε όλο τον εθνικό τους. Για να δούμε επομένω τι μορφή θα πρέπει να λάβουν οι προπολογισμοί και πώς μπορούν επίσης οι εθνικοί προπολογισμοί να πρασινίσουν περισσότερο με αυτούς τους ε, μίνιμουμ στόχους δαπανών εν ώψη του πλαισίου για το 2030. Για δούμε τώρα τι γίνεται με την προστάμινη ενωσιακή ε, αξία και αυτόν τον ελάχιστο στόχο. Είναι σημαντική η αύξηση των δαπανών για το κλίμα. Μίλαμε για 180 δις ευρώ το 2011 και τώρα έχουμε 200, πάνω από 200 τέλο δις 7% στην προηγούμενη περίοδο, για τον προηγούμενο προπολογισμό, αλλά και για τα διαρθρωτικά επιδικά ταμεία, η χρηματοδότηση από το 12% πήγε στο 21%. Άρα, αυτή η αύξηση στις δαπάνες και η συμπερίληψη του θέματος σε όλες τις πολιτικές σημαίνει ότι ο στόχος έχει προσθεμένη αξία και άρα θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και για το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Πρέπει επομένως να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Τώρα, να δούμε εντάχει αυτό. Έχω εδώ πέρα από το 2017. Βασική τομή δαπανών. ΚΑΠ 27% για την ε, πολιτική συνοχή, 7% το Horizon 2020, 1% το Life και το Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία. Και 10% οι λοιποί τομεί. Όπω προαναφέρθηκε, μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα σε άλλου τομεί. Ασφάλεια, ιδιώτες πολίτη, κοινωνικό ταμείο κλπ. Τώρα, διαζόμαστε από το χρόνο, οπότε πάμε λίγο πιο γρήγορα, παρακάτω. Άρχισε κανεί μια ματιά σε αυτά τα ποσά, αυτέ τις δαπάνες, διαφορετικές χρονιές και έχουμε ε, τώρα για την προβολή, την πρόγνω, το προγνωστικό του για το 18-20, βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει χρόνο να αναλυφθεί η δράση. Παρ' όλα αυτά η προσδοκία δεν είναι το να φτάσουν το 20% στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο πήραμε αλλά δεν πρέπει να φτάσουν σε κορεσμό. Γιατί από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατόν να πάει 20% για το κλίμα. Οπότε τα προγράμματα δράσης και θα μια διεξοδική αξιολόγηση του ποια πολιτική πώς μπορεί να βοηθήσει μέχρι 20%. Χρειάζεται να γίνει αυτό. Τώρα, βελτίωση στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων. Το Ελληνικό Συνέδριο το, το είπε και η τράπεζα ότι έχουμε αυτό τον συντελεστή του 100% που αφορά τη Συμφωνία του ΡΙΟ τους σχετικούς δείκτες. Αυτό να αφορά το, σημαντικό κομμάτι. Αλλά υπάρχει και το 40% που είναι πιο περιορισμένης σημασίας. Να πώς γίνεται η διάθεση των δαπανών ε, όταν είναι οι δείκτες λιγότερο αυστηροί από τα όσα επιτάσσει ο ΣΑΚ. Έτσι έχουμε υπερεκτίμηση των δαπανών. Αυτά για το tracking, αυτά για τις εκθέσεις. Σε σχέση με τα προγράμματα δράσης που είπαμε όσον αφορά τις αιτήσεις εκθέσεις, για τη χρηματοδότηση και για επί τη βάση της τι θα πρέπει να γίνει τώρα. Όσον αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ποσά των δαπανών αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις ε, επιπτώσεις όσον αφορά την προσπάθεια για το κλίμα. Οπότε θα μπορούσαμε να προτείνουμε να υποβάλλονται εκθέσεις ε, εκ των προτέρων και των υστέρων ε, όσον αφορά τις ε, εξοικονομήσεις σε εκπομπές ή τις εκπομπές για τα αέρια του θερμοκηπίου. Πόσα τέτοια σώζουμε και πόσο πόσα εκπέμπονται. Γιατί Έχουμε έκθεση για την ΚΑΠ, έχουμε για το Περιφερειακό Αναπτυσιακό Ταμείο και για το ορίζον 2020 δεν έχουμε σχετική έκθεση. Άρα θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε για όλους τους τομείς όπου προβλέπονται δαπάνες. Τώρα, εδώ να δούμε τα έχει. Έπειτα έχουμε χρόνο το ότι υπάρχει κάποιο είδους έλλειμμα στον αυτό τι, τι, τι αξιοποιούν οι 13 τα ταμεία για τι δαπάνε. Ε, οι 13 είναι το γκρι και οι υπόλοιποι είναι το πράσινο. Άρα και εδώ μπορούν να γίνουν ε, βελτιώσει. Τώρα, όσον αφορά την αναβάθμιση του προγράμματο live, την ενίσχυσή του, αυτό θα πρέπει να μελετηθεί διότι όσον αφορά το κλίμα ε, ε, ε, είναι 100% το πρόγραμμα. Και για κάθε 100 ευρώ όλα πάνε στο κλίμα και όχι 25. Και το 25 ευρώ ή λιγότερο. Και βλέπουμε ότι και εδώ όσον αφορά το πρόγραμμα για την ευφύ ενέργεια θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μελετήσει κατά πόσον ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να ε, αναπρικοδοτηθεί γιατί ξεκίνησε με μόνο 500 εκατομμύρια και αυτό σχέση με το 2020 θα μπορούσε να αυξήσει την χρηματοδότηση. Επομένως βλέπουμε ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες με ε, τους στόχους για 2050 και θα πρέπει να συνεχιστούν οι δαπάνες οι ελάχιστε κλιματικές δαπάνε, θα πρέπει να υπάρξει στεγανή παρακολούθηση και υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Ε, θα πρέπει επίσης να ε, κάνουμε στεγανή την, ε, την νομοθεσία για τα αποτυπώματα του άνθρακα και οι 13 θα πρέπει να βοηθηθούν και επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τα προγράμματα που είναι 100% κλιματικά. Merci. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, διακόπτω και σας πιέζω. Ε, ε, ο καθένας θα λάβει γνώση του εγγράφου και θα κανονίσει την πορεία του. Τώρα το λόγο έχει ο δεύτερος εμπειρογνώμων του πάνελ, ο κύριος Έρο Γύριο Κόσκινεν, διευθυντής του Green Budget Europe. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αξιότιμη και εκλεκτή προσκεκλημένη. Είναι τιμή για μένα να έχω ε, την ευκαιρία να παρουσιάζω ε, στην παρούσα συνεδρίαση ε, την απόψή μας. Το Green Budget Europe είναι μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στους περιβαλλοντικούς φόρους και άλλα εργαλεία της αγοράς για να μειωθεί η επιβλαβής δράση στο περιβάλλον. Ανθρωπογενής θα βασιστώ σε δύο προηγούμενες εκθέσεις μας, μία του 2016 που αφορούσε τους ιδίους πόρους, γιατί τους πράσινους και ε, το δεύτερο φορά τους φόρους, ε, τους πράσινους, πάλι η έκθεση του 2016. Θα αρχίσω την παρουσίαση αυτή εξετάζοντας ε, το παρόν σύστημα ιδίων πόρων. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, η σημαντική ε, πλειονότητα του προπολογισμού προέρχεται από εθνικές συνεισφορές de facto. Το μεγαλύτερο μερίδιο ε, είναι ένα ποσοστό του ΟΕΠ ή διάφοροι πόροι. Αυτό που οδήγησε στην ε, ενιαύσια δημοσιονομική διαδικασία υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο ενώ η κανονική πανευρωπαϊκή στάση και συμπεριφορά ε, παραγνωρίζεται και κάθε χώρα ε, αγωνίζεται για τη δίκαιη επιστροφή των χρημάτων της. Le juste retour λέγεται αυτό στα γαλλικά, ε, που δεν είναι πάρα πολύ ευβίωνο για τη μελλοντική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άρα θα ήταν μάλλον φυσικό να θεωρήσει κανείς ότι χρειάζεται προσπάθεια διαφοροποίησης ε, των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σταδιακή μετάβαση σε γνήσιους ιδίους πόρους. Πράγμα που θα αυξήσει και το ρόλο του Κοινοβουλίου αλλά ε, και θα το θεωρεί και η ιδιοκτησία του ε, αυτό ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης. Απότερο στόχος πιστεύω ειλικρινά ότι θα είναι να καταρτίζεται ένας ουσιαστικά αυθεντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με διπλά ωφέλη. Πέρα από τις κλασικές χρηματοδοτήσεις ε, των πολιτικών μας, βεβαίως θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στις διεθνείς μας υποσχέσεις για την ανάπτυξη γενικά, για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της βλάβης στο περιβάλλον. Από τις δύο λοιπόν αυτές εκθέσεις που σας ανέφερα του 2016 εντοπίσαμε ορισμένες επιλογές για ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων που αναγράφονται όπως βλέπετε στις διαφάνειες, φορολόγηση των καυσίμων των οδικών μεταφορών, φορολόγηση διοξιδίου του άνθρακα, άλλοι ενεργειακοί φόροι, πράσινα δασμοί ε, και ε, ε, φόρο στα πλαστικά και τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη φορολόγηση των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές. Οι οδικές μεταφορές, ε, είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς, αποτελούν τον μοναδικό κλάδο ε, στις μεταφορές όπου αυξάνονται τα αέρια του ε, θερμοκηπίου. Επίσης είναι και η βασική υπέτη για την ατμοσφαιρική ρήπανση που είναι ολέθρια για την ανθρώπινη υγεία. Και σε πολλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές των καυσίμων των οδικών μεταφορών, πράγμα που προκαλεί και μεγάλες ε, στρεβλώσει στον ανταγωνισμό. Μπορεί να έχετε ακουστά ε, τον ε, τουρισμό για λόγους καυσίμων, για να βάλει κανείς καύσιμα σε άλλη χώρα. Επίση είναι πολύ σημαντικές κάποιε εξωτερικές παράμετροι, δηλαδή πώς επηρεάζει ο τομέας των μεταφορών, όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη συμφόρηση, την κυκλοφοριακή. Ε, η φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα θα έχει στόχο να δημιουργήσει ίσους κανόνες παιχνιδιού με ένα βασικό συντελεστή ε, φορολόγησης εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα που δεν καλύπτεται από το σημερινό σύστημα του πρασινίσματος. Αυτό τι θα έδειχνε. Πρώτον ότι είναι προσιλωμένη στους στόχους του ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη Συμφωνία των Παρισίων και θα έπρεπε να στρέψει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές σε νέες μορφές ενέργειας χαμηλής παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα. Ένας ενεργειακός φόρος θα μπορούσε να είναι η αύξηση στο περιεχόμενο της ενέργειας και όχι στον όγκο που δεν συμβαίνει σήμερα. Ας πούμε η φορολογική αντιμετώπιση του άνθρακα. Ε, είναι πολύ χαμηλή, ενώ θα πρέπει να είναι υψηλότερη. Και έχουμε και τους νέους στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Ε, στη συνέχεια, οι πράσινοι λεγόμενοι δασμοί επίσης είναι μια επιλογή ενδεχόμενη. Αυτό θα ήταν μια προσαρμογή στα σύνορα ε, ως προς το διεξίδιο του άνθρακα για να αντισταθμιστούν κάποιες ε, πλεονεκτικές τιμές που έχουν ε, χώρες που παράγουν ε, κάποια αγαθά ε, με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και έρχονται και τα πολλούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Μοιραία είναι φθηνότερα όλα αυτά. Μήπως χρειάζεται να αντισταθμιστεί στα σύνορα αυτό ως πράσινος δασμός που θα επιβάλλεται έτσι ώστε να συνάδουν καλύτερα οι εμπορικοί με τους περιβαλλοντικούς μας κανόνες. Επίσης, τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ίδιος πόρο Βεβαίω βεβαίως αυτό το σύστημα έχει ένα πλεονέκτημα γιατί ήδη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα μπορούσε να επαναπροσανατολιστεί για να χρηματοδοτήσει κάποιες δραστηριότητες. θα είπε και ο ε, προλαλής σας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες. Η μία του κυρίου Έτιγκερ, του Επιτρόπου, για το φόρο στα πλαστικά, στις πλαστικές σακούλες. Αυτό το κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εξετάζουν και στον Ηνωμένο Βασίλειο και άλλο Υπουργείο Οικονομικό. Βεβαίω ο φόρο στα πλαστικά δεν θα είναι βασική πηγή χρηματοδότησης των ιδίων πόρων, αλλά συμπληρωματική προς άλλες υφιστάμενες. Συνεχίζουμε. Σε κάποιες συστάσεις θα ήθελα να περάσω τώρα. Πρώτον, εμείς πιστεύουμε ότι όλες οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να συνάδουν με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ε, επίσης, η οριζόντια εγκάρση στόχη αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη στις τρεις βασικές ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, κοινή γεωργική πολιτική, διαρθρωτικά ταμεία και το επόμενο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Εκτός αυτού βεβαίως θα ήταν φρόνιμο και θα συνιστούσαμε να μπουν νέοι ήδη διπόροι, με αυτούς τους περιβαλλοντικούς φόρους να ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους στόχους που έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας και να δίνουν ένα πολιτικό μήνυμα στα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και να τους καθοδηγούμε προς την κατεύθυνση που στοχεύουμε. Και τέλος, για να συνοψίσω κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αξίζει να επανέλθουμε και να δούμε ποια είναι η σημερινή κατανάλωση ενέργειας, πώς διαφρόνεται αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε ο Επίτροπος Άριας Κανιέτε πριν από 15 μέρες, κατά 72% η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, απορρικτά καύσιμα. Έχουμε δεσμευτεί όμως εμείς με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και αυτό το ποσοστό θα πρέπει να μειωθεί και να φτάσει σχεδόν στο μηδέν μέχρι το 2050. Αν θέλουμε να ε, συμμορφωθούμε με τη Συμφωνία των Παρισίων. Άρα κύριε Πρόεδρε είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε στο στόχο αυτό εκτός εάν ε, εισάγουμε νέα ε, υποστηρικτικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Κάποιο είδου φορολογική μεταρρύθμιση θα χρειαστεί ή εργαλεία που να βασίζονται στην αγορά για να οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ήθελα να σας δείξω κι άλλα πώς κατανέμεται η κατανάλωση ενέργειας στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα, που είναι οι δύο χώρες που παράγουν τα περισσότερα ε, αέρια του θερμοκηπίου. Δεν έχω αυτή την κατανομή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον επιμερισμό. Θα ήταν όμως ενδιαφέρον το δούμε, γιατί θα μας ανοίξει τα μάτια. Εδώ βλέπουμε όλη τη δομή της ενεργειακής κατανάλωσης στις Ηνωμένε Πολιτείες και μετά έχουμε κόψει εκεί μια φέτα που δείχνει ε, την ηλεκτρική ενέργεια και τον επιμερισμό αυτής της συγκεκριμένης ενέργειας ε, στην κατανάλωση. Εκεί είναι μεγαλύτερες επιδόσεις και τα επιτέγματα. Εκεί αυξάνεται το μερίδιο των ανανεωσίμων και αυτά κυριαρχούν στις ειδήσει. Αλλά μόλις 20% είναι η ηλεκτρική ενέργεια, και από ανανεώσιμες. Όλα τα υπόλοιπα, μεταφορές, θέρμανση, βιομηχανική παραγωγή, όλα αυτά βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα που θα πρέπει να ξεφορτωθούμε στα επόμενα 30 χρόνια, που είναι μικρό διάστημα. Είναι μεγάλη η πρόκληση και δεν πρόκειται να γίνει με τους σημερινούς μηχανισμούς. Απλούστατα αυτό που μας χρειάζεται είναι νέα κίνητρα και όχι μόνο και άλλα μέτρα για να έχουμε μαζικές επενδύσεις στις νέες υποδομές και αντισταθμιστικά μέτρα για να καλυφθούν οι απώλειες των θέσεων εργασίας. Υπό την έννοια αυτή η ήδη πόροι πράσινοι θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί για την μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια πιο πράσινη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Πολύ ανησυχητική εικόνα. Διότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι γιγαντιαίου μεγέθους. Και ατυχώς βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν για την εκείνη τη προς επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων. Euh, Έχει κάποιε ερωτήσεις. Όποιο θέλει, μιλήσει τώρα. Ε, λακωνικότατη παρακαλώ. κυρία Τόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχόλιο. Έχοντας ακούσει τους εμπειρογνώμονές μας, συμφωνώ με αυτό που είπατε κύριε Πρόεδρε απηχεί και την τελευταία παρέμβαση. Στην πραγματικότητα είμαστε μηδαμινοί σε αυτή την ιστορία. 1% του ΑΕΠ, ο προπολογισμό της Ένωσης, ενώ θα χρειαζόμασταν ίσως να το τετραπλασιάσουμε, πενταπλασιάσουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να είμαστε αποτελεσματικοί. Το λέω εκ του προχείρου. Εγώ θα τηρήσω αυτά που έγραψα στην έκθεσή μα. 1,3 όριο, οροφή. Πρέπει να είμαστε πραγματιστέ, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι γελίο. Γελίο σε σχέση με το διακύβευμα. Είπαμε να πάμε 4% των δαπανών υπέρ του κλίματος. Θέλουμε να συγκλίνουν οι πολιτικές συνοχής γεωργίας προς το κλίμα. Καλά θα ήταν όλα αυτά όσον αφορά τις επιδόσεις, να είμαστε καλύτεροι. Αλλά αν δεν υπάρχει σχέδιο μεγάλων επενδύσεων, δεν θα ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα τα κάνουμε όλα καλά, θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και σχέση με το 30% που ψηφίσαμε που δεν θέλει να ακολουθήσει από ό,τι βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαστε στεναροί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό άκουσα και εξέλαβα από τις παρεμβάσεις εκτός αν σφάλω, θα χρειαζόμασταν πολλαπλασιασμό του προπολογισμού. Θέλουμε τετραπλάσιο, πενταπλάσιο προπολογισμό της. Ε, δεν ξέρω, από αυτά που είπατε, γνωρίζετε ότι θα έπρεπε να κάνουμε το Συμβούλιο. Ότι Um, Θα είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Uh, Κύριε Σέφα, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα LIFE και τη συνεισφορά του, που είναι αποκλειστικά για το περιβάλλον και τη βιοπικιλιότητα κάποιοι ΕΣΜΙΚΙΟ εντόπισαν κάποια δυνατότητα που έχει το ΛΑΕΦ. 1% του προπολογισμού της ΑΕΠ για αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνοντας το Natura 2000 κλπ. Ρεαλιστικό είναι αυτό το επίπεδο. Ποιο θα ήταν το ρεαλιστικό επίπεδο για αυτό το πρόγραμμα, διότι το 0,3% που έχουμε είναι προφανώς ανεπαρκές. Δεν υπάρχει άλλος που να ζητάει το λόγο. Πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Τωμά, θέλει τετραπλάσιο, πενταπλάσιο προϋπολογισμό. Μπορούμε να φανταστούμε το δεχόμενο κάποιες δαπάνες που αναλαμβάνονται από τα κάτι μέλη σε επίπεδο εθνικό για το κλίμα, των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν είναι βέλτιστη. Διότι για να έχουμε αποτελεσματικότητα πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέω, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια φορά αυτές οι δαπάνες από εθνικό επίπεδο να περάσουν σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μειωθεί η δημόσια δαπάνη σε εθνικό επίπεδο και να αυξηθεί η δημόσια δαπάνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας για την προστασία από τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος και για την προστασία του περιβάλλοντος. Καλό τους δύο πυρογνώμονες να απαντήσουν στις παρατηρήσεις που έγιναν. Παρακαλώ όσο πιο σύντομα μπορείτε. Um, um, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σέφερ, για τις ερωτήσεις σας. Και... Βέβαια, και είναι μικρή φέτα από το ΑΕΠ. Αλλά θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε σε σχέση με το Brexit πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και από πού θα προέλθουν τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσπάθησα να σας πω στην προσοχή μου είναι το εξή. Η Ένωση είναι το πράγμα προς για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αρκετά λεφτά στον προπολογισμό. Και αν ναι, τι γίνονται. Πώς θα χρησιμοποιούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι σαν ανάλυση κόστους ε, αποτελέσματος και να δούμε πόσες σε ε, εκπομπές αερίων θερμακηπίου μπορούν να ξεκονομηθούν, να κοπούν να μειωθούν ανά ευρώ και έτσι κανείς να κάτσει και να δει τι γίνεται με τα προγράμματα, της πρωτοβουλίας, τι αποδίδουν και ποιο αποδίδει περισσότερο και φυσικά θα ήταν επιθυμητό να ήταν πιο πλούσιος ο προπολογισμό και να μπορούσε να κάνει περισσότερα. Αλλά πολλά μπορούν να γίνουν με ό,τι υπάρχει. Και κανείς να καθοδηγήσει τα κράτη-μέλη πώς μπορούν να πρασίνσουν τους εθνικούς προπολογισμούς, οπότε κανείς καταλήγει στον ίδιο λογαριασμό που δαπανάται. Βέβαια, μπορεί κανείς να μετακινήσει τους πόρους, να μεταφέρει πόρους από τα κρατημέλη προς τον κοινωνικό προϋπολογισμό, το οποίο βέβαια είναι πολιτικό θέμα και μέχρι ποιο άμα θέλουν τα κρατημέλη έτσι να αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύουν στον κοινωνικό προπολογισμό. Και αυτό χωρί συζήτηση. Ποιο θα ήταν το σωστό ποσό για το live. Δύσκολο το ερώτημα. Κάνει θα πρέπει να δει το live μέχρι ποιο βαθμό έχει ξεπεράσει τους τεθέντες στόχους για το κλίμα. Να το δει αυτό ποσοστία και σύστηχα να αυξήσει τη χρηματοδότηση. Ε, πάντως δεν είναι και σημαντικά τα σχετικά ποσά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το τι θα αποτελούσε επαρκές ποσό αύξησης. Αλλά σα είπα και αυτά τα, για αυτά τα προγράμματα στην πρόσθεση μου ότι για κάθε ευρώ που αυξάνηκαν στον προπολογισμό τότε πάμε στο 100% πάνε αυτά τα, τα, τα λεφτά δηλαδή τη αύξηση στο κλίμα το οποίο δεν ισχύει για τα περισσότερα άλλα προγράμματα που αφορούν άλλου τομεί. Για αυτά τα προγράμματα κάθε ευρώ πάει ολόκληρο στο κλίμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κόσκινεν. εθνικοί προπολογισμοί και κοινοτικοί στόχοι. Ε, είναι το θέμα λεπτό. Αλλά αν δούμε τις διαφορετικές εναλλακτικέ, όπως σας τα είπα, καταλήγουμε ότι η καλύτερη υποψήφη κορυφή θα ήταν το εισόδημα του ETS, ε η ενεργειακή φόρη. Βέβαια, το πρόβλημα με τους φόρους επί της ενέργειας είναι ότι προς το παρόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εθνικού εισοδήματος από τους φόρους. Και πάντως μία από τις ε, δικαιολογίες θα ήταν ότι η αλλαγή του κλίματος δεν γνωρίζει σύνορα. Και θα υπήρχε προστιθέμενη αξία εάν κάποια από αυτά τα χρήματα πηγαίνανε σε κοινωνικούς στόχους. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα ολοκληρώνουμε την ακρόαση και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας που μας διαφώτισαν. Ήταν εξαιρετική ποιότητα τα όσα μας είπατε. Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε. Οπότε να, αυτά όλα αφορούν τη Συμφωνία των Παρισίων. Και περιμένουμε να ακούσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτές και για τους νέους ιδίους πόρους. Συμφωνούμε όλοι και αυτός είναι ο λόγος που κάναμε την κοινή ακρόαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Το πρόβλημα για το κλίμα είναι μείζον πρόκληση που αφορά τον πλανήτη, τη ζωή, την ανθρωπότητα. Και ακριβώς όπως ελέγχεται στο τέλος μπορούμε να συνδέσουμε το ζήτημα των ίδιων πόρων με τις δαπάνες διότι για να μπορούμε να λάβουμε δράση όσον αφορά την νοοτροπία μας θα πρέπει να συνδυαστούν τα μεν τα δε. Και δεν μπορώ να ξεχάσω την ομάδα ψηφοπαίδου του Μόντι που έλεγε ότι το σωστό είναι να υπάρχει ένα κονδύλι για το κλίμα στον προπολογισμό της Ένωση. Και ε, βλέπουμε τι γίνεται με πόρους, δαπάνες, δημόσιες δαπάνες, δαπάνες των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων, όλων όσοι θα πρέπει αλληλέγγυα να φροντίζουν για την μείωση των εκπομπών. ενωπιστων των στόχων 2030-2050. Οπότε παραμένει περιορισμένο το προϋπολογισμό προπολογισμό μας, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις πιστώσεις που έχουμε, τους πόρους που έχουμε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε το tracking και το reporting γιατί θα πρέπει για τα προγράμματα να μπορούμε ε, ξεκάθαρα να δούμε ποια είναι τα αξιόλογα στοιχεία, αυτά τα οποία μας δείχνουν αποτελεσματικότητα κλπ. Να μπορούμε να, να υπολογίσουμε την ευρωπαϊκή προστιμένη αξία, γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος και οι φορολογούμενοι. Δηλαδή να ρίχνουμε στον προπολογισμό χρήματα και να προκύπτει όμως προς θεμένη αξία. Επίσης, θα πρέπει από αυτούς τους λίγους πόρους που έχουμε να βρίσκουμε κάτι για να πιέζουμε τα κράτη-μέλη, τους οικονομικούς ε, παράγοντες, τους ε, πολίτες, με τις δημοσίες δαπάνες, όχι με κυρώσεις, αλλά με την φορολογική τους εισφορά. Να κάτσουμε μέσα να προβληματιστούμε με αυτές τις ενδιαφέρουσες και πολλά υποσχομένες ακροάσεις. Τώρα όμως, για να ολοκληρώσω, θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τάραντ, που δεν εγκατέλειψε ούτε δευτερόλεπτο το έδρανό του. Σας ακούμε. Uh, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα συνοψίσατε άριστα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που ξόδεψαν τον πολύτιμο χρόνο τους εδώ. Συνοψίζοντας, τα παιδιά μου που είναι ευρωσκεπτικιστές με ρωτάνε «Μα τι κάνετε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο αν δεν μπορεί να αλλάξετε κάτι» και να τους δώσω παρηγοριά τους λέω, είναι σαν τα μεταπτυχιακά. Εκεί μπορείς να συναντήσεις ε, ταλεντούχους ανθρώπους, έμπειρους, να σου δώσουν συμβουλές και να σε σπρώξουν στο πολιτικό σου πρόγραμμα μέχρι το πικρό τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur Taran. Ευχαριστώ κύριε Ταρόν. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω ότι θα συνεχίσετε να επαγρυπνείτε. Και η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θα προβεί στις αξιολογήσεις με αυστηρότητα και συνέπεια. Ιδού ευχαριστώ τους επαΐοντες, ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ρέλ και τον κύριο Όεν και έχουμε την ελπίδα ότι στις 2 Μαΐου θα έχουμε μια επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ότι ήταν καλύτερο για να προστατεύσει το κλίμα. Θα διακόψουμε τις εργασίες μας και καλώ τους συναδέλφους να μετακινηθούν στην PHS 4Β 01 011 για το εξωτικό σχέδιο επενδύσεων μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ναι. Euh, Ευχαριστώ λοιπόν και τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Διακόπτεται η συνεδρίαση.